Très bien. Je, je vais vous proposer de, de démarrer nos, nos travaux. Si vous voulez bien. Euh... Je dois tout d'abord euh, excuser le président. Να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του Προέδρου, ο οποίος δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σήμερα. Τουλάχιστον όχι στην αρχή. Θα έρθει λίγο πιο μετά. Και έτσι λοιπόν ε, θα προεδρεύσω εγώ προς το παρόν ε, των εργασιών της Επιτροπής μας. Μου ζητήθηκε να τον αντικαταστήσω στην αρχή της συνεδρίασης. Με μεγάλη μου χαρά. Να εγκρίνουμε λοιπόν καταρχάς την ημερήσια διαδάξη. στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης, η κυρία Γκέρλινγκ. Θα θέλαμε να αποσύρουμε αυτή την έκθεση, να την αναβάλουμε προς, να την αναβάλουμε για τις 7 και 8 Νοεμβρίου και να αντικατασταθεί το σημείο αυτό από την παρουσίαση από την DG Santo της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των θεμάτων για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Αυτά. Αυτή είναι η μοναδική τροποποίηση που έχω να προτείνω για τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε αντίληση, θα ήθελα να θεωρήσω την ημερήσια διάταξη εγκεκριμένη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Θα σας ενημερώσω ότι η συνεδρίαση μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο με το web streaming και επίσης έχουμε διερμηνία σε 16 γλώσσες για σήμερα και αύριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρακτικά της συνεδρίασης της 30 Αυγούστου, δεν λάβαμε οποιαδήποτε ένσταση αντίρρηση σε ό,τι αφορά τα πρακτικά αυτά, άρα θεωρούνται εγκεκριμένα, εφόσον δεν έχετε καμία αντίρρηση. Πολύ ωραία. Εγκρίνονται. Και έτσι περνάμε στο πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Και θα ζητήσουμε από την ε, συνάδελφό μας τη Μαρία Νόχη να μας κάνει μια πρώτη παρουσίαση των θέσεων για το σημαντικό αυτό θέμα της συγκέντρωσης των ε, γεών και το πώς θα διευκολυνθεί η πρόσβαση στην γη για τους γεκτήμονες, για τους αγρότες. Η Μαρία λοιπόν είναι η συγκεντριά μας και θα πάρει το λόγο για μια πρώτη ανταλλαγή άποψε. για να κάνουμε μια πρώτη ανάλυση του θέματος αυτού. Η γη, καταλαβαίνετε, είναι η βάση της γερικής παραγωγής. Και τίθεται το θέμα, λοιπόν, των εκτάσεων αυτών. Έχουμε τα θέματα του και τα θέματα των πλημμυρών, τα θέματα τα πολιτισμικά, όλες αυτές οι διαστάσεις ε, συνδέονται με τις εκτάσεις αυτές. Και σε κάποιες ε, φάσεις, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και το θέμα της ε, χρήσης του όρου, της χρήσης ή της εγκατάλειψης της γης όταν πρόκειται για ορεινές περιοχές και το καθεξής. Η κερδοσκοπία σε ολόκληρη την Ευρώπη οδηγεί σε μεγάλη συγκέντρωση των γεών και εμποδίζει την πρόσβαση για τους ε, μικρούς ε, γεωκτήμονες. Αυτό το παρατηρούμε σε όλα τα κράτη-μέλη για μια ισότιμη πρόσβαση στις γης για την οικονομική γεωργία σε μικρή και μεσαία κλίμακα. Ε, χρειαζόμαστε νέα δυναμική στην Ήπεθρο και νέες προϋποθέσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας είναι ε, κέρια σημασία, διότι και κάνουμε τώρα την ενδιάμεση αναθεώρηση, αλλά και επεξεργαζόμαστε τι κατευθυντήριε γραμμέ ε, για την πολιτική μετά το 2020. Έτσι, θα έχουμε τα νέα μέσα για να θέσουμε αμφιβόλο την ε, τρέχουσα ανάπτυξη και να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει σε ευρωπαϊκή κλίμακα και να αντιμετωπίσουμε το μεγεθυνόμενο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι γεωργοί αλλά και οι οργανισμοί ανάπτυξη τη υπαίθρου καθώς ε, και όλες ε, οι ενώσεις ε, στην επικράτεια των κρατών μελών που δρούν και αγωνίζονται για αυτά τα σκοπό. Ελπίζουμε να κάνει συγκεκριμένε προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτόν τον τομέα στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του γεωργικού κόσμου στην Ευρώπη. Δεν θέλω να παρατείνω την εισαγωγική μου παρουσίαση. Σας δίνω το λόγο, θα κάνετε την αρχική παρουσίαση και μετά θα γίνει ανταλλαγή απόψεων και φυσικά μετά θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Νόησλη. Ganz herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender, für das Wort. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα καταρχά. Είναι το πρώτο θέμα αυτό στην ημερήσια κατάκτηση σήμερα το πρωί, το θέμα τη κατάσταση σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση των χερσαίων γεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η δυνατότητα απόκτηση πρόσβαση ε, στι ε, καλλιεργήσιμε αυτέ εκτάσει. Πρόκειται για μία έκθεση πρωτοβουλία, δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι σε κενό αέρο που αναπτύχθηκε αυτή η πρωτοβουλία. Υπήρχε μία παρόμοια το 2014 με τίτλο Άγρα χερσαίων γέων σε ό,τι αφορά τις οικογενειακές ε, επιχειρήσεις. Ήταν μια έκταση η οποία εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία στην Οικονομική και Γεωργική ε, Επιτροπή Γεωργικής Ανάπτυξης και το 2014 είχαμε το θέμα του land grabbing στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε και μια αναφορά για το θέμα αυτό, για το τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το φαινόμενο αυτό. Παγκόσμια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αυξάνεται δηλαδή η συγκέντρωση των χερσαίων γεών. Αυτό απειλεί ασφαλώς τις επιχειρήσεις, τι μικρές, τις οικογενειακές, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά, αν θέλετε, και το, της παραγωγής και ε, της ε, καλής διαχείρισης της γης. Κάποιες τώρα σκέψεις να σας παρουσιάσω. Πρώτες σκέψεις σήμερα, τα οποία, τις οποίες τις έχω αναφέρει και τις έχω γράψει και στο έγγραφό μου και θα ήθελα να συζητήσουμε μετά. Έχουμε λοιπόν τα στοιχεία, τα δεδομένα επιτάπητα στο 2010. 3% των επιχειρήσεων παρέγαν 50, είχαν μάλλον 50% του μεριδίου των γεών των καλλιεργήσιμων. 3% δηλαδή των επιχειρήσεων ελέγχουν το 50% των εκτάσεων και 18% 80% ε, έχουν μόνο 14,5% των γεών. Και αυτό. Και στη Βραζιλία, στην Κολομβία και στις Φιλιππίνες ισχύει ε, κάτι τέτοιο. Αλλά Κοιτάξτε, εμεί ε, στην Ευρώπη ήμασταν περήφανοι γιατί θεωρούσαμε ότι είχαμε καλύτερε αναλογίε και καλύτερε ισορροπίε, αλλά διαπιστώνουμε ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τι χώρε αυτέ. Land grabbing τώρα. Αυτό το. η των γιών. Αυτό το κατηγορούμε και το επικρίνουμε σε ό,τι αφορά τις ε, φτωχές ε, χώρε υπερβολική δηλαδή συγκέντρωση των γεών. πώ είναι δυνατόν να μαζεύεται όλο και πιο μεγάλες εκτάσεις σε όλο και λιγότερα χέρια. Θα ήθελα και το τονίζω αυτό στην έκθεσή μου ότι δεν είναι εμπορεύσιμο αγαθό και μεταβιβάσιμο αγαθό η γη και δεν είναι και απεριόριστο χωρίς ε, περιορισμούς το αγαθό αυτό. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, λοιπόν, θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσον η αργή τη ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου, την οποία φυσικά και την διατηρούμε στην Ευρώπη, κατά πόσο μπορεί να ισχύσει λοιπόν και για τις καλλιεργήσιμες αυτές εκτάσεις και φυσικά αυτό συνδέεται και με την προσδοκία για κέρδος, αυτό διακρίνει και οδηγεί σε κερδοσκοπία, αλλά οι προσδοκίε των ομίλων είναι διαφορετικέ από τι προσδοκίε του πολίτη και του καταναλωτή, ο οποίο θέλει α, τρόφιμα, βιοενέργεια, σε ό,τι αφορά τι πρώτε τα κτλ. Άρα οι εκτάσει η γη γίνεται όλο και πιο ακριβή. Αλλά δεν αυξάνεται φυσικά σε ποσότητα και αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις. 2007-2008 ξεκίνησε ιδιαίτερα αυτή η φαρπαγή γεών. Τότε που ξεκίνησε και η οικονομική κρίση και η κρίση της πείνας ε, στην, ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η γη λοιπόν δίνει δυνατότητα παραγωγής ενέργειας, παραγωγής τροφίμων. Και εδώ πραγματικά βλέπουμε μια μεγάλη τέτοια τάση στην παρούσα φάση. Φυσικά υπάρχουν και παράνομε δραστηριότητε και διαδικασίες στην Ευρώπη. Πέρα από τα τελωνία δηλαδή, λένε ότι τη μεγαλύτερη ε, διαφθορά λαμβάνει χώρα σε θέματα μεταβίβασης και χρήσης της γης. Μεγάλος τομέας λοιπόν που διακρίνεται από ιδιαίτερη διαφθορά και ο κίνδυνος που φυσικά προκύπτει από τη συγκέντρωση γεών, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι και τι πρόβλημα υπάρχει που συγκεντρώνονται σε λίγα χέρια η γη και οι εκτάσεις ίσα ίσα. Θα μπορούσε να είναι και θετικό για την παραγωγή τροφή μόνο. Αλλά αυτό δεν ισχύει, ξέρετε, σε καμία περίπτωση. Γιατί το θέμα της ιδιοκτησίας και της κατοχής ε, εκτάσεων και της εκμετάλλευσης και της ιδιοκτησίας ε, διαχωρίζεται και δημιουργείται ένα χάσμα μεταξύ των δύο αυτών ενιών. Για παράδειγμα, στην Σλοβακία έχουμε 96% μίσθωσης εκμίσθωσης υγεών. Και αυτή η μεγάλη συγκέντρωση των υγεών προκύπτει από διάφορα ζητήματα. Δεν υπάρχουν δηλαδή επενδυτές, επενδυτέ που αγοράζουν, μάλλον υπάρχουν μεγαλοεπενδυτές που αγοράζουν μεγάλες εκτάσεις για να κερδοσκοπήσουν. Δεν έχουν πραγματικά συγκεκριμένη σύνδεση με την καλλιέργεια. Υπάρχουν και ε, διαδικασίες αγοράς ε, από μεγάλους ομίλους που έχουν ως σκοπό συγκεκριμένη καλλιεργία και θέλουν ουσιαστικά να αυξήσουν το μέγεθος των ομήλων τους. Αυτές οι αγορές λοιπόν στην εσωτερική, στο εσωτερικό της Ευρώπης ε, μάλλον αυτέ οι, μεγάλοι όμιλοι ε, προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλέ περιπτώσει, αλλά και εκτό Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως για παράδειγμα οι Κινέζοι οι οποίοι συχνά καταφέρνουν και αγοράζουν yes, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσο μπορούμε να αντιτηρήσουμε το βιώσιμο μοντέλο καλλιέργεια, το οποίο χαρακτηρίζεται από τι οικογενειακέ επιχειρήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η συγκέντρωση γεών εξαρτάται και διακυβεύει το πώς ε, ορίζουμε την ε, κατοχή και την διεκτησία γεών. Το θέμα της κατανομής ε, Τη ιδιοκτησία των γεών έχει να κάνει και με την κοινωνική ασφάλεια, με τον κοινωνικό ιστό, με την εσωτερική ασφάλεια, αν θέλετε, των κρατών. Και η συγκέντρωση των γεών, και εδώ υπάρχουν μεγάλες έρευνες που μπορείτε να διαβάσετε, οδηγεί λοιπόν σε μη αναστρέψιμες ζημιές στον κοινωνικό ιστό. Οδηγεί μικρές πόλεις, κομμοπόλεις και χωριά στην αναδιάρθρωση της ίδιας τους, της σύνδεσής τους. Αλλάζει η γονιμότητα του εδάφους, αλλάζει η παραγωγή τροφίμων και αυτό συνεπάγεται ε, μειονεκτήματα, όχι μόνο για την Ήπεθρο, αλλά και για την ίδια τη γη. Και απειλούνται φυσικά και ιδιαίτερως οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, γιατί αυτοί παράγουν το μεγαλύτερο τμήμα των ε, τροφίμων, των βιώσιμων τροφίμων, των ε, α, υγιεινών τροφίμων. Δεν μιλάμε μόνο για την επισητιστική ασφάλεια, αλλά μιλάμε και για αυτή την πολυτροπική γεωργία, την οποία έχουμε θέσει στο επίκεντρο των προτεραιότητων μας. Εγώ πιστεύω και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τον τίτλο. Ο τίτλος της έκθεσης καταδεικνύει ότι αφενός θέλουμε να βάλουμε στο επίκεντρο την παρουσίαση των ε, γεγονότων, των αριθμητικών στοιχείων και θα πρέπει να καθορίσουμε και τις προτεραιότητές μας. Λοιπόν, η προτεραιότητα θα πρέπει να τεθεί από τους πολιτικούς ευθύνοντες και θα πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα διαμορφωθεί η πολιτική ε, εδαφούς μέσω της ε, στρατηγικής μας για τη συγκέντρωση υγεών. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή χώρες να περνάνε νομοθεσία για την προστασία των γεών του, για να μην υπάρχει συγκεντρωσή στα κέρια μεγάλων και από την άλλη να βρίσκονται σε μηνυτική θέση και να του απειλεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν επιτρέπεται να το κάνουν αυτό. Γιατί αν η γη α, ανήκει αποκλειστικά στα κράτη-μέλη και είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, δεν θα πρέπει να επιτρέπονται Διαδικασίε παρέμβαση και επίσης χρειαζόμαστε και σαφή κριτήρια στη τελική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πότε και τι μπορεί να κάνει μια χώρα για να προστατεύσει τις καλλιεργέσιμε εκτάσει τη. Και είναι σημαντικό λοιπόν οι χώρες να μπορούν να περνούν και τη νομοθεσία. Για παράδειγμα, ανώτατα όρια για την ιδιοκτησία, για την ενεργή ε, αγορά γεών για την χρήση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων από τόπιους και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί. Χρειαζόμαστε σαφήνεια τι επιτρέπεται να κάνει μια χώρα για να προστατεύσει την γη της. Και έτσι λοιπόν μας λείπουν και πάρα πολλά δεδομένα. Δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή διαμόρφωση της κατάστασης, μια ευρωπαϊκή επισκόπηση για το ποιο έχει τι μερίδιο των γεών. Κατεπηγόντως χρειάζεται αυτό. Και μια τελευταία σκέψη, επιτρέψτε μου. Η πολιτική μας ε, για την γεωργική πολιτική, για τις επιδοτήσεις στα πρωτοπυλώνα. Αναφέρει ότι, μάλλον ε, θέτει σε αμφισβήτηση μεγάλο τμήμα της ε, πολιτικής για τη γεωργική ανάπτυξη. Όταν λοιπόν σας λέω ότι 3% των επιχειρήσεων κατέχουν 50% των ε, εκτάσεων, ε, εδώ τίθεται το θέμα των επιδοτήσεων. Και έτσι με τη σειρά του, αυτέ οι επιχειρήσει. το 3% αγοράζει ακόμα πιο πολύ γη. Και έτσι ουσιαστικά η πολιτική και οι επιδοτήσει τη γεωργική πολιτική συνεχίζουν αυτή την τάση συγκέντρωση. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε παρατηρητήρια, θα πρέπει να καταγράψουμε επακριβώ την κατάσταση και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να υπάρχουν και θελούσιε κατευθυντηρίες γραμμές για την ε, ανάπτυξη για την εκμετάλλευση των καλλιεργήσεων γεών. Και θα πρέπει να είναι πιο υποχρεωτική αυτή η παρουσίαση των δεδομένων για να ξέρουμε πώς μπορούμε και πώς παρεμβαίνουμε στην πολιτική αυτή. Γιατί η πρόσβαση στη γη είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Και για να επανέλθουμε και στον τίτλο της έκθεσης, σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση των, των γεών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε όλα αυτά αν απλοποιήσουμε την κατάσταση. Αν οι καλλιεργήσιμες γέες παραμένουν σε λογικές τιμές, γιατί όταν οι τιμές φτάνουν σε μη ρεαλιστικά επίπεδα, πώς θα έχουν οι αγρότες πρόσβαση στη, στη γη. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα συζητήσουμε και ευχαρίστως να κάνουμε μια πολύ ζωηρή συζήτηση και φυσικά εάν έχετε σχόλια και παρατηρήσεις ευχαρίστως να τα στείλετε στο γραφείο μου. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή θα αποτελέσει μία βάση η οποία θα χρειαστεί και ενώπιον της νέας μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, η οποία κάποια στιγμή θα είναι αναπόφευκτη. Και θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τη σύνδεση με την αποτροπή της συγκέντρωσης των χερσαίων γιών. Ευχαριστώ, Μαρία, για αυτή την εισαγωγική παρέμβαση θέτει στο πλαίσιο της συζήτηση. Πολύ ζητήσατε το λόγο. Η ημερήσια διάταξη όμως είναι επιβαρημένη. Θα έλεγα λοιπόν 1,5 λεπτό ο καθένας. Θα ξεκινήσω με τους κοιόδης εισηγητές. Για 1,5 λεπτό πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Μαρία. Και εγώ πιστεύω ότι η γη είναι ένα κοινό αγαθό, την οποία θα πρέπει να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ως προτεραιότητα την παραγωγή τροφίμων. Νομίζω ότι και η απόδοση και η αγορά ε, για τους αγρότες θα πρέπει να είναι δυνατή. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μηχανισμούς για να ε, εμποδίσουμε τις απαλωτριώσεις, ε, την εγκατάλειψη των γεών κτλ. Δεν θα πρέπει να αλλάζουμε τη χρήση της γεωργικής γης επίσης. Θα πρέπει να έχουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς. Επίσης, να διευκολύνουμε την πρόσβαση για τους νέους και για τα άτομα που θέλουν να εγκατασταθούν, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επίσης να δώσουμε ειδική προσοχή στην πρόσβαση ε, από γυναίκε στη γη. Νομίζω ότι θα πρέπει να απαγορεύσουμε και τελειώνω γιατί δεν έχω χρόνο καταστάσεις υφαρπαγής ε, γόνιμων γεών μέσω απαλωτριώσεων ε, και είναι συχνά οι πρώτες γέες που εξαφανίζονται, οι πιο γόνιμες δηλαδή, ε, καθώς και πρακτικές γεωργικές οι οποίες ε, θίγουν την ε, ικανότητα παραγωγής ε, τροφίμων από διάφορα από τις γέες και την πλήττουν, ας πούμε, με τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η έκθεση για αυτό το θέμα, γιατί αυτό το θέμα είναι θέμα κεφαλαιόδου σημασία. Δεν είναι μόνο η βάση για τους γεωργούς, Νομίζω ότι είναι ε, η βάση της ζωής για όλους. Και είναι και το μέλλον μας. Ό,τι καταστρέφουμε σήμερα θα το πληρώσουν οι επόμενες γενιές επίσης. Το είπε η Μαρία. Η γη δεν είναι ένα αγαθό όπως οποιοδήποτε άλλο. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα όμως. Κυκλοφορεί πολύ χρήματα, πολύ χρήμα. Οι χρηματαγορές δεν, ψάχνουν, δεν μπορούν να βρουν κάτι ενδιαφέρον για να επενδύσουν και αγοράζουν λοιπόν γη όσοι έχουν λεφτά. Τη, τη γη τη θεωρούμε ως ε, περιουσιακό αγαθό, ε, την αντιμετωπίζουμε ως ε, εμπορεύσιμο είδος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μπει στη γωνία της, ας πούμε, και να πει ότι τα θέματα αυτά είναι εθνικής κυριαρχίας. Ναι, είναι. Αλλά θα πρέπει ως Ευρώπη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλουμε κάποια ορόσημα. Έχουμε νομοθεσία και δεν μπορεί να τη χρησιμοποιούμε μόνο για να παρεμβαίνουμε, μόνο να παρεμβαίνουμε στην εσωτερική αγορά και στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Πρόκειται για θεμελιώδη θέματα. Υπάρχει το θέμα της διαφάνειας, υπάρχει το δικαίωμα που έχουν ε, οι γεωργοί να έχουν γη για να την εκμεταλλευτούν και πρέπει να υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο στις ε, τιμές της γης γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν ποτέ να αγοράσουν οι γεωργοί. Νομίζω ότι αυτές οι κατευθυντήριες, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να εφαρμοστούν και στην Ευρώπη και θα πρέπει να ορίσουμε το είδος γεωργίας που επιθυμούμε. Παρακαλώ να σας υπενθυμίσω ότι έχετε 1,5 λεπτό ο καθένας. Επιτρέψτε μου να σας το υπενθυμίσω, γιατί αλλιώς δεν θα καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε την ημερήσια διάταξη. Η κυρία Μιούλερ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Μαρία Νόεχλ που μας έκανε αυτή τη διεξοδική παρουσίαση, περιέγραψε με ακρίβεια την κατάσταση και επίσης ε, θεωρώ ότι ε, σε αυτό το τομέα των επενδύτων ε, θα πρέπει να δράσουμε, δεν μας μένει τίποτε άλλο, ασκείται μεγάλη πίεση σε αυτές τις μικρές γεωργικές επιχειρήσεις. Επίσης, χαιρετίζω το ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλουμε να υιοθετήσουμε μια κοινή προσέγγιση. Θα ήθελα λοιπόν να ενισχυθεί αυτή η τάση. Ε, χωλένουμε ως προς την πολιτική σε σχέση με το έδαφος και του, της ΓΕΣ. στην ε, Γερμανία υπάρχουν τρία διαφορετικοί νόμοι για την ενίσχυση των μικρών γεωργικών επιχειρήσεων ε, και την ενίσχυση της ενεργού γεωργίας. Δυστυχώς στην πραγματικότητα συμβαίνουν άλλα πράγματα. Ε, υπάρχουν ε, επίσης από την Επιτροπή του ΙΕ ε, κατευθυντήριες γραμμές προαιρετικές για την ασφάλεια στον τομέα της διαχείρισης των γεών. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις εκμισθούμενες γεές, διότι με τις επιδοτήσεις ενισχύουμε αυτή την αρνητική τάση ε, σίγουρα θα υποβάλω τροπολογίες ε, για να προσθέσουμε ενδεχομένως σε κάποια σημεία ε, κάποια άλλα στοιχεία. Σας ευχαριστούμε. Ε, Σκιώδης για το ΕΛΚ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νόχιλ, διότι ήγερε τα σημαντικά ζητήματα που θα συζητήσουμε σήμερα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι γεύσεις είναι η βασική ε, πηγή τροφίμων και άρα δεν μπορούμε να τη μεταχειριζόμαστε ως οποιοδήποτε αγαθό είναι περιορισμένο, πόρος και ε, εξασφαλίζει την επιστημιστική ασφάλεια. Γι' αυτό και πιστεύω πως θα πρέπει να διαφυλάξουμε την ποιότητα των οικογενειακών γεών και να εξασφαλίσουμε πρόσβαση για αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονται. Μικρή γεωργή, παραγωγή, δηλαδή και ενεργή γεωργή. Θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω κάποιε που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει η έκθεση. Πρώτον, ορισμός της συγκέντρωσης των γεών. Τι σημαίνει αυτό. Ε, θα πρέπει να κάνουμε διάκριση σε σχέση με άλλες διαδικασίες, όπως αυτό που ονομάζουμε land consolidation. Ε, ε, δηλαδή, αυτό μπορεί να είναι καλό κατά τη διαστολή με τον κατακαιρματισμό των υγειών, Ενοποίηση, λοιπόν, μικρών γεωτεμαχίων. Θα πρέπει, λοιπόν, να αναρωτηθούμε η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ποιο βαθμό ε, ενθαρρύνει ή παρεμποδίζει την πρόσβαση στη, στα αγροτεμάχια. Σε ποιο βαθμό οι επιδοτήσεις ε, ενισχύουν τα μεγάλα επενδυτικά ταμεία, ε, σε ποιο βαθμό τα μέτρα που αναλαμβάνουμε προστατεύουν ε, τους μικρούς γεωργούς. σε πληροφορίες για την ε, μεταβίβαση ε, γεών δεν υπάρχουν και γι' αυτό θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Καλή επιτυχία κυρία Νόηση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βοπέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. εξαιρετικά επίκαιρο αυτό το ζήτημα. Μαρία, σε ευχαριστώ που ανέλαβες αυτό το μοιράκλειο έργο. Ε, η Υπάρχει στην εθνική αρμοδιότητα. Όμως εμείς θα πρέπει να προσδιορίσουμε τις κατευθύνσει τη κοινή γεωργικής πολιτική. Μέσα από του υποστηρικτικούς μηχανισμούς λοιπόν τη κοινή γεωργικής Πολιτική. θα πρέπει να έχουμε κάποιες δικλείδε ασφαλείας για να αποφύγουμε καταστάσεις όπως παραδείγματος χάρη την κερδοσκοπία που γίνεται σε βάρος των γεωργών. Ε, τις επιδοτήσεις μας σε διάφορους γεωργικούς τομείς, σε ποιο μέγεθος ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να τις κατευθύνουμε, γιατί αυτό πρέπει να αποφύγουμε, δηλαδή να μην αγοράζονται, να μην εξαγοράζονται υγιές μόνο και μόνο για τις επιδοτήσεις κοινή γεωργικής πολιτικής. Επίσης, ε, να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας. Ποιος θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ε, το ε, αγροτεμάχιο. Ε, στη Λιθουανία, παραδείγματος χάρη, έχει προτεραιότητα ο γείτονας. Εάν δεν θέλεις να πουλήσεις το αγροτεμάχιο στο γείτονά σου, τότε αρχίζουν να ισχύουν άλλα, άλλες διατάξεις. Ευχαριστώ. Κύριος ε, Λοζό. Ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ την ε, εισηγήτρια. Η συγκέντρωση των αγροτεμαχίων και των εκμεταλλεύσεων όντω είναι ένα πραγματικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήστε που είναι και ουσιαστική απειλή ε, κατά της παραδοσιακής γεωργίας ε, σε ε, χώρες Ανατολικής Ευρώπης, στη Ρουμανία παραδείγματο χάρη, ξένα κεφάλαια αγοράζουν τα αγροτεμάχια και οι γεωργοί υποφέρουν από την φτώχεια, δεν έχουν πρόσβαση στα αγροτεμάχια, αλλά αυτέ τι τάσει παρατηρούνται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί η επιφάνεια των αγροτεμαχίων κατά 38% κατά μέσο όρο και ο κατακαιρματισμό είναι ο μεγαλύτερος ε, στην Ευρώπη, στη Ρουμανία ε, και 20 με 30% ε, των επενδυτών στην Ευρώπη έχουν το μεγαλύτερο αριθμό αγροτεμαχίων, το ίδιο και στην Βουλγαρία παραδείγματο χάρη στην Πολωνία. Μόνο 1% των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων ελέγχουν το 20% των ε, αγροτεμαχίων στην Ευρώπη, όπως είπατε, και 3% το 50% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ε, αυτό δημιουργεί ανισορροπία και ε, δυσχεραίνει την πρόσβαση στα αγροτεμάχια για τους ε, γεωργούς. Ε, είναι αυτή η διγλωσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που τελικά υπονομεύει την παραδοσιακή γεωργία και ενισχύει την βιομηχανική γεωργία μέσω της συγκέντρωσης των γεων. Αυτή η υπερφιλελεύθερη πολιτική σας το μόνο που κάνει είναι να οδηγεί σε υπερσυγκέντρωση των γεών. Θέλω να έχουν ανθρώπινο μέγεθος οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις Όλα απολούνται, όλα αγοράζονται σε αυτόν τον νεοφιλελεύθερο κόσμο. Ποια μέτρα εσείς θα αναλάβετε για να καταπολεμήσετε την κερδοσκοπία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Μαρία μίλησε για ένα διπλό κίνδυνο. Και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τις πολιτικές μας. Καταρχάς, να χάσουμε τις γεωργικές γεές και να υπάρξει μια αστικοποίηση και να ε, εξαφανιστούν τα δάση. Επίσης υπάρχει πρόβλημα ε, υπερμεγέθυνσης, ευτροφισμού των εκμεταλλεύσεων που θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στον γεωργικό κόσμο και κυρίως στην απασχόληση. Για το θέμα τη ε, της κληρονομιάς επίσης πρέπει να το δούμε γιατί είναι τεράστιο θέμα. Ε, κληρονομιά ε, ήδη μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας είναι περίπλοκο γιατί υπάρχουν ε, αδερφοί και αδερφές που δεν έχουν τις ίδιες ιδέες για τη γεωργία. Ε, υπάρχουν και χειρότερα όμως. Ε, κληρονομιές εκτός οικογένειας που πλέον δεν γίνεται, δεν υπάρχει λόγω του κόστους ε, της γεωργικής γης. Όταν ήμουν πρόεδρος περιφερειάρχης είχα βάλει μία διάταξη ε, ούτως ώστε να υπάρχει μία δυνατότητα μίσθωσης. Δηλαδή η περιφέρεια με τη βοήθεια του ΦΕΝΤΕΡ ε, αγόραζε κάποιες γεωργικές γεές, τις ε, αποθήκευε ούτως ώστε να μπορούν να εγκαθίστανται οι νέοι γεωργοί εκεί. Τους τις νίκιασε σε πρώτη φάση, εν συνεχεία τις κληρονομούσαν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να βρούμε μηχανισμούς ούτως ώστε να, να κρατήσουμε την ε, γεωργική δραστηριότητα στα ανθρώπινα μέτρα ε, ο γεωργός της γειτονιάς να μπορέσει να ασκήσει το επάγγελμα αυτό και όχι να έρθουν οι ξένοι επενδυτές. Νομίζω ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε την απόλυτη ανάγκη να διατηρήσουμε τον έλεγχο στην ε, γεωργική γη και οι δημόσιες αρχές και η Ευρώπη να παίξουν ένα ρόλο εκεί. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα της ιδιοκτησίας της γης δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, μην το ξεχνάμε. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δω την Ευρωπαϊκή Ένωση να χώνει τα, τη μύτη της στην ιδιοκτησία της γης. Είναι τέλειο το σύστημα, έχουμε ένα κτηματολόγιο εμείς και πολύ εύκολα μπορούμε να δούμε ποιος, σε ποιο ανήκει τι. Υπάρχει αίσθηση ότι το μικρό είναι τόσο όμορφο και το μεγάλο είναι άθλιο ε, σας παρακαλώ. Ε, για κοιτάξτε ε, τι γίνεται σε μια φυτή, ας πούμε, ε, πώς γίνεται, τι χρησιμοποιούμε τώρα, ας πούμε, με τις μεγάλες μηχανές και 30 α, χρόνια πριν. πριν από 40 χρόνια είχαμε τον απλό ας πούμε τον εργαζόμενο ο οποίος προσπαθούσε να μόνος του να μαζέψει ας πούμε τα ζαχαρότεφλα ας πούμε ε, που αρουρέει παντού κτλ. Ενώ σήμερα έχουμε τεράστια ωραία μηχανήματα κτλ. Ε, και τι να κάνουμε. Χρειαζόμαστε λιγα, λιγότερους ανθρώπους ε, σήμερα. Ο πατέρας μου το 1948 ας πούμε ήθελε πολύ περισσότερους ας πούμε. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε συνέχεια το ρολόι πίσω. Τι προσπαθεί να πετύχει εδώ η συγγήτρια. Προσπαθεί να πετύχει να μας πει ότι τόσοι θα είναι ας πούμε ε, στη γη και θα τους πληρώνουμε δεν και καλά ότι και δουλεύουν δεν δουλεύουν ας πούμε με τα λεφτά των φορολογούμενων ας πούμε μια εθνικοποίηση της γης, μια κοινωνική πολιτική ή λέτε ότι θα πρέπει να αναδιοργανώσουμε την διοκτησία της γης ούτως ώστε το περιβάλλον να βελτιωθεί. Κι όμως δίνουμε, ας πούμε, ε, πληρώνουμε ας πούμε, για να εξασφαλίσουμε την ε, ποιότητα και του νερού και της γης κτλ. Και δεν έχει σημασία ποιο είναι ο ιδιοκτήτης. Είναι το άτομο ας πούμε, το οποίο φροντίζει αυτή τη γη, ο οποίος παίρνει αυτά τα λεφτά ούτως ώστε να εξασφαλίσει την ε, ποιότητα της γης. Δεν χρειάζεται να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς για να το πετύχει αυτό. Τι πράγματα είναι αυτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήμουν υπέρ του να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα η γη να καταλήγει στα χέρια των ε, αγροτών που θέλουν να την καλλιεργήσουν. Είτε είναι μικροί καλλιεργητές, είτε είναι μεγάλη όμιλη. Και θεωρώ ότι έτσι θα δώσουμε μια διάσταση στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Αλλά να αναφέρω και ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στην Κροατία. Η κροατική κυβέρνηση από το 2000 μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να διαχειριστεί σωστά την γεωργική πολιτική, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κρατικές, τις δημόσιες yes. Έχουμε λοιπόν... Έχουμε λοιπόν τη Σλαβωνία με, με τεράστιες εκτάσεις, όπου το κράτος θέλει να προστατεύσει τα δημόσια συμφέροντα, αλλά έχουμε και μικρές ε, ολορίδες γεών στις παράκτιες περιοχές όπου ο κόσμος θα ήθελε να έχει ιδιοκτησία των εκτάσεων αυτών και να καλλιεργεί, για παράδειγμα, ελιές. Άρα, στην Κροατία, ο κόσμος θέλει να έχει στην κατοχή του την ιδιοκτησία του γη, αλλά τα δυσκολεύεται πράγματα η κυβέρνηση. Είναι πραγματικά παράλογη αυτή η πολιτική. Άρα εγώ θα ήθελα να έχουμε κατευθυντήριες γραμμέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μας κατευθύνουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χόισλινγκ. Χόσλινγκ. Σας ευχαριστούμε κυρία Νόχιλ για την ε, έκταση. Να τη δούμε κιόλα. Αλλά θεωρώ ότι τα ευρωπαϊκά αριθμητικά στοιχεία είναι ε, απαραίτητα να τα έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί ενδιαφέρει η κατάσταση φυσικά. Και στη Γερμανία την ίδια. Διαφέρει η κατάσταση στην Ανατολική Αποτεβητική Γερμανία, πρώην Ανατολική Αποτεβητική. Γιατί φυσικά υπήρχαν και διαφορετικές ιστορικές ε, συνθήκε. Άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε τα πράγματα πιο συγκεκριμένα. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε τι δυνατότητε έχουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα δεν είναι μόνο η κατανομή των ε, γεωργικών μέσων. Το θέμα είναι και κατά πόσον ε, η καταποκοπή επιδότηση ουσιαστικά ευνοεί τις μεγάλους ομίλους, γιατί βλέπουμε ταχύτερη ανάπτυξη των μεγάλων ομίλων από ότι των μικρών επιχειρήσεων. Άρα ουσιαστικά αλλάζει η αναλογία και ευνοούνται οι μεγάλοι όμιλοι. Και να δούμε λοιπόν όλες αυτές οι πολιτικές που ακολουθούμε, πόσο ωφελούν τους μεν και τους δε. Θα πρέπει επίσης να το εξετάσουμε και είναι σημαντικό αυτό. Θα πρέπει να καταφέρουμε επιχειρήσεις που δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με την γεωργία και απλά θέλουν να επενδύσουν ε, στην γεωργική εκμετάλλευση να βγουν εκτός παιχνιδιού. Δεν είναι δυνατόν να είναι δηλαδή οι ιδιοκτήτε εταιρείε οι οποίε να έχουν, έχουν μόνο το κεφάλαιο και να μην ασχολούνται καθόλου με την καλλιέργεια. Αυτό θα πρέπει να το αποτρέψουμε πάση Ευχαριστώ. Ο κύριος τόρφμαν Σας ευχαριστώ. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και με τα στατιστικά στοιχεία, να δείξουμε λίγη προσοχή, γιατί τα στατιστικά στοιχεία έχουν πάντα λίγο υποκειμενική αξία και θα πρέπει να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Υπάρχουν, για παράδειγμα, μέρη στην Ευρώπη, όπως τις ε, Νότιες Άλπης όπου υπάρχει αντίθετο πρόβλημα. Μπορώ να σας πω, για παράδειγμα, τυχαίνει και ένα εκτάριο να έχει 20 διεκτήτες. Και αυτό στο παρελθόν είχε οδηγήσει σε τόσο μεγάλο κατακαιρματισμό της διεκτησίας των γεών και οδήγησε σε προβλήματα στην αγορά. Η συγκέντρωση λοιπόν θα ήταν πάρα πολύ θετική και ευπρόσδεκτη στις περιοχές αυτές και θα ήθελα να επαναλάβω και σε αυτά που είπε ο συναδελφός Χόισλινγκ. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτούμε κατά πόσον η πολιτική μας και οι επιδοτήσεις στον πρώτο πυλώνα ουσιαστικά προωθούν λαθασμένες καταστάσεις. Και αυτό γίνεται, πιστεύω. Οι εξελίξεις ε, στην ε, πολιτική, μάλλον, ήταν διαφορετικές στο παρελθόν πλέον ε, από ότι είναι πλέον σε, σε συνθήκες ε, κρίσης. Και ενδεχομένω να έχουν αλλάξει κάποια ώρες τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Είναι ε, εκεί που συμφωνώ με την κυρία Νόιχλ είναι το, στο εξή. Θα πρέπει να δώσουμε στα κρατή-μέλη τη δυνατότητα να αποφασίζουν τα ίδια το πώς ε, κληροδοτείται η γη, πώ πωλείται η γη. Αυτό που δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουμε. Να, είναι να επιτρέψουμε, αυτό που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνουμε, είναι να επιβάλλουμε ε, κάποια ανισορροπία μέσα στα κρατημέλη, τα οποία για κάποιο λόγο έχουν αποφασίσει να περάσουν μια συγκεκριμένη νομοθεσία σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία. Θα πρέπει να ισχύουν ήδη όροι για όλους, ακόμα και σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία και την κατοχή υγεών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στές. Να τονίσουμε λοιπόν κάποια στοιχεία, γιατί σε κάποια με βρίσκω, είμαι σύμφωνο, σε κάποια άλλα έχω κάποια ερωτηματικά. Άρα, ε, είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ, υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ καταστάσει, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην ίδια Γερμανία μέσα. Από τη Βαυαρία είμαι, θα το ξέρετε, και ε, η μέση έκταση διοκτησιών είναι 15-16 εκτάρια στην περιοχή μου. Δεν πωλείται η γη. είναι σπάνιο φαινόμενο και έτσι δεν έχουμε πρόβλημα κατανομής ε, και διασκορπισμού. Το θέμα φυσικά της μίσθωσης και τα λοιπά έχει να κάνει με τη διάρθρωση της γεωργίας. Και πριν από κάποιο α, καιρό ήμουν στην Ανατολική Γερμανία όπου είναι τεράστια η συγκέντρωση αλλά και εδώ θα πρέπει να κάνουμε διάκριση για παράδειγμα μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν ενδεχομένω 261 ιδιοκτήτε, αλλά σε κάποιε περιπτώσει μιλάμε για επιχειρήσει ε, που έχουν 350 εκτάρια και άλλοι είναι υπεύθυνοι για το οικονομικό σκέλος και άλλοι είναι υπεύθυνοι για την καλλιέργεια. Είναι πολλά και διαφορετικά λοιπόν τα μοντέλα. Και να μην ξεχνάμε και το θέμα, για παράδειγμα, της οικοδόμησης υποδομών, οι οποίες ε, αποστερούν μεγάλο μερίδιο των καλλιεργήσιμων γεών και θεωρώ ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή εδώ και να δούμε και τι γίνεται με την ιδιοκτησία της γης γενικότερα. Ευχαριστώ κύριε Σουφάναγκανο. Thank um, Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας, ε, κυρία Νόιτσελ. Αναρωτιόμαστε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να τη διευκολύνει τη συγκέντρωση των γιών. Ε, και τι εννοώ. Ε, ε, μπορεί ένας γεωργός να πάρει χίλια ευρώ για ένα εκτάρι και ο γείτονας τίποτα. Ε, ή έρχονται και παίρνουν μισό εκατομμύριο ευρώ. Ε, ε, ενώ οι ανταγωνιστές τους δεν παίρνουν τίποτα. Ε, οι μεγαλογιοκτήμονες δηλαδή παίρνουν όλες τις επιδοτήσεις. Ε, μπορούμε λοιπόν να κάνουμε αυτό που πρότεινε ο τελευταίος αξιοπρεπής επίτροπος, να έχουμε ένα front-loaded σύστημα με ανώτατο όριο πληρωμών μπορούμε να το κάνουμε αυτό κατά την αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Δυστυχώς όμως ο τωρινός επίτροπος, ο κ. Χόγκεν, δεν υποστηρίζει αυτή την ιδέα. Ε, και ακούω πράγματα που με ξαφνιάζουν. Βλέπω ότι υπάρχει υποστήριξη για τις μικρές εκμεταλλεύσεις, ακόμη και από το ΕΛΚΑ. Όταν ναι, επιλέξαμε λοιπόν τον Επίτροπο, εγώ αντιτάχθηκα στο Χόγκαν ναι, γιατί ε, θεωρούσα ότι δεν θα υποστηρίξει αυτή την ιδέα, όχι γιατί σε τοπικό επίπεδο ε, ήταν ανθυποψήφιος, ε, αλλά διότι θεωρούσα ότι δεν θα υποστήριζε αυτή την ιδέα και θα πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο επιτρέπει επιλέξαμε αυτόν τον επίτροπο που υποστηρίζει την αγριοβιομηχανία και όχι τους ε, μικρούς ε, ε, γεωργούς. Έρχεται λοιπόν ο μεγαλογεωκτήμονας και πετάει με ελικόπτερα και παίρνει τις επιδοτήσεις ενώ αυτοί που θα έπρεπε να παίρνουν τις επιδοτήσεις δεν έχουν λεφτά ούτε για να βάλουν ντίζελ στο τρακτέρ. Ευχαριστούμε κύριε Φλάνακαν. Ο κύριος Βούντα. Ευχαριστώ. την ε, κυρία Νόεχλ ε, για την ε, παρουσίασή της. Θέλω να καταγγείλω την υποκρισία της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέει, είναι ανησυχητικό αυτό το φαινόμενο που επεκτείνει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη μας λέει ότι πρέπει να το λύσουν το πρόβλημα τα κράτη-μέλη. Εγώ μπορώ να σας πω ότι στη Ρουμανία προσπαθήσαμε να τροποποιήσουμε την νομοθεσία για την ε, μεταπόληση μεγάλων αγροτεμαχίων. Ε, δεν μπορούσαμε ε, να το κάνουμε, να υλοποιήσουμε την ιδέα γιατί δεν μας άφησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα αυτά λέμε ισχύει ε, ισότιμη πρόσβαση στα αγροτεμάχια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπω ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε νομοθετικό επίπεδο για την πώληση υγειών στα κράτη-μέλη ε, τη Ευρωπαϊκή Νομίζω δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει στην πράξη. 47% των υγειών στη Ρουμανία είναι στα χέρια ε, ξένων ε, επενδυτών. 45%. Οι πρώτες δέκα εταιρείε ως προς τον αριθμό των επιδοτήσεων είναι από το Λίβανο, από όποια χώρα μπορείτε να φανταστείτε. Σίγουρα όχι από κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, εάν και αυτό δεν θα μας ενοχλούσε αν όντως ε, υπήρχε μια παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Αλλά αυτές οι μεγάλες εταιρείες ούτε καν ε, ε, διατηρούν την ποιότητα του εδάφους. Εγκαταλείπουν αυτά τα τεμάχια και μόνο παίρνουν τις επιδοτήσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να παθήσουμε να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Κατεπηγόντως θα πρέπει να επιβάλλουμε εναρμονισμένες διατάξεις για την πόλη των γεών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κύριος ε, ευχαριστώ. Μαρία, νομίζω ότι γενικά επικρατεί εντύπωση στην Επιτροπή. Έφυγε ο Άντριο. Α, εδώ είσαι. Ε, ο Στιούαρτ ε, ε, ανήκει στη μειοψηφία. Η πλειοψηφική άποψη στην Επιτροπή είναι ότι όντω υπάρχει πρόβλημα και Στιούαρτ υπάρχει και μια τροχιά εδώ που διαγράφεται. Αν ε, λοιπόν συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο σε πέντε χρόνια θα δεις ε, δει ότι το 2% των εκμεταλλεύσεων θα έχουν το 75% των ε, γεών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Νομίζω ότι για όσους είναι ε, στην αριστερά ε, ε, αποδεικνύει την αποτυχία της αγοράς. Δύσκολα θα το παραδεχτεί το ΕΛΚ. Δεν λειτουργεί σωστά η αγορά και βλέπουμε ότι διευρύνεται το χάσμα, οι, φτωχότεροι, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι και συγκεντρώνεται η γη σε λιγοστά χέρια, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτή είναι η γενικότερη εικόνα. Δείτε το ειδικτυσιακό καθεστώς στο Λονδίνο ενώ οι αλλοδαποί ιδιοκτήτες, ε, ε, λίγοι ε, στον αριθμό, κατέχουν τις περισσότερες, τα περισσότερα κίνητα. Ε, τώρα, ε, ε, η αλλαγή στο σύστημα των πληρωμών είναι μία από τις πιθανές λύσεις στην Ουαλία. Ε, ισχύει ήδη το ανώτατο όριο, όχι στη Σκωτία, όχι στην Αγγλία, στην Ουαλία. Και αυτό εφαρμόζεται σε τρεις μόνο γεωργούς, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα ανώτατο όριο. Είναι λοιπόν μία πιθανή στρατηγική για να σημειωθεί η πρόοδος. Νομίζω ότι είναι μια λύση που θα πρέπει να εξετάσουμε και ποια είναι η πράξη, ε, τι συμβαίνει στην πράξη, ε, χρησιμοποιούνται οι επιδοτήσεις ε, εις βάρος της γεωργίας και αυτός δεν, είναι, δεν ήταν ο στόχος της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστούμε πολύ, ο Τζέιμις Νίκολς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και στην Ιρλανδία το κάνουμε αυτό. Βάζουμε ανώτατο όριο δηλαδή στην τιμή της γης όχι μόνο στην Ουαλία. Πάντως, ε, δεν υπάρχει πια γη που παράγει φρούτα, ας πούμε. Ε, όλο και λιγότεροι είναι, ε, την, την τσιμεντώνουν, σηκώνουν α, ψηλά κτίρια, σπίτια, εργοστάσια, οτιδήποτε. Άκουσε το νούμερο του 3% και του 50%. Νομίζω ότι πρέπει να τα ψάξουμε αυτά τα νούμερα περισσότερο. Γιατί θα ήθελα να ξέρω πού συμβαίνουν αυτά. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα της συγχώνευσης, ας πούμε, γεών ε, σε κάποιες ε, νέες ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε κάποιες παλιές. Πάντως, Νομίζω ότι η μία λύση που καλύπτει κάθε πραγματικότητα ε, δεν είναι σωστή για την Ευρώπη. Στη δική μου περιοχή, όταν είχαμε την οικονομική ανάπτυξη, είχαμε δικηγόρους, ε, είχαμε αρχιτέκτονες, ε, ερχόντουσαν ας πούμε, στην πόλη μας ας πούμε, και αγόραζαν μικρούς λοφίσκους και έχτιζαν σπίτια κτλ. Σταμάτησαν όλα αυτά. Το πρόβλημα με εμά είναι ότι οι τράπεζες στην πραγματικότητα μπαίναν μπροστά ας πούμε και δώσαν, δίνανε δάνεια σε όλους όσους θέλαν να αγοράσουν γη γιατί το θεωρούσαν τεράστια και πολύ καλή επένδυση. Μερικές φορές μου λένε οι αγρότες ότι δεν βγάζουν λεφτά. Το θέμα είναι να δούμε ποιο έχει τα λεφτά. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ποιο έχει τα λεφτά για να αγοράσει τη γη. Ο κύριο Μπόγκοβιτ. Ευχαριστώ Μαρία για την έκθεση αυτή. Πολύ σημαντικό το θέμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε. Είμαι Σλοβαίνος ένα γεωργό κατά μέσο όρο έχει 6,7 εκτάρια. Μερικές φορές χρειάζεται η συγκέντρωση, ούτω ώστε οι νέοι γεωργοί, οι μεσαίοι γεωργοί να μπορούν να βγάζουν τα προστοζήνα από αυτή την ε, γεωργική εκμετάλλευση. Στις ε, πρώην κομμουνιστικές χώρες είχαμε μεγάλα κομμάτια, μεγάλα τεμάχια δημόσιας γης, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ε, γιατί συχνά πέρασαν στα χέρια ενός ιδιοκτήτη και είναι λάθος αυτό. Είναι πολιτική, ας πούμε, η φαρπαγή της γης. Γιατί προτιμούμε την ε, γεωργία η οποία βασίζεται σε μικρές εκμεταλλεύσεις, σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Έτσι πρέπει να δούμε αυτό το πρόβλημα της υφαρπαγής της γης. Από την άλλη να προετοιμάσουμε και μέτρα για να υποστηρίξουμε κυρίως νέους ε, γεωργούς και μεσαίους μεσαίας κλίμακας γεωργούς για να οργανώσουν τη γεωργική τους εκμετάλλευση με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν και να ζουν από αυτή τη γη. Θα πρέπει λοιπόν επίσης να έχουμε και διαφορετικά μέτρα για διαφορετικές χώρες, γιατί δεν είναι παντού η κατάσταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Κόστιντζερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να συνεχίζω τη σκέψη που ξεκίνησε ο συνάδελφο. Αυτό που είναι καθοριστικό και θα είναι καθοριστικό να το διευκρινίσουμε στην έκθεση είναι ότι η αρμοδιότητα είναι στα χέρια των κρατών μελών και ότι και ανακάρτω μέλος τα πράγματα διαμορφώνονται διαφορετικά αναπεριφέρεια, αναμόσπονδο κρατήδιο, γιατί για παράδειγμα στην Αυστρία έχουμε πολλέ διαφορέ. Πρώτα γεγονό ότι είναι μικρή χώρα, ιστορικός πω. ήταν διαφορετική η πρόοδος, η εξέλιξη σε ό,τι αφορά το θέμα των κληροδοτημάτων, σε ό,τι αφορά το θέμα της κληροδότησης των γεών. Όλα αυτά λοιπόν αφορούν ιδιαίτερα τους νέους γεωργούς που κληρονομούν, οι οποίοι είναι και πολύ πιο επιτυχείς, αν θέλετε, πολύ πιο οικονομικά αναπτυγμένοι σε περιοχές της Αυστρίας που υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία για τη συγκέντρωση των γεών από τις άλλες περιοχές όπου τα πράγματα είναι πολύ πιο κατακαιρματισμένα και είναι πιο, πιο δύσκολη η οικονομική αξιοποίηση. Και θα πρέπει να λάβουμε λοιπόν υπόψη ότι είναι διαφορετικές οι καταστάσεις ένα κράτος μέλος, ότι αυτό είναι θέμα αρμοδοτήτων των κρατών μελών και ότι διαμορφώνται διαφορετικά καταστάσεις και μέσα στα κράτη-μέλη. Να βρούμε και διατυπώσεις οι οποίες στο μέλλον και στο μέλλον ε, θα αποτρέψουν καταστάσεις όπου θα πηγαίνει κάποιος ιδιοκτήτης να αγοράσει υγιές σε ένα κράτος μέλος, ένα σολοδαπός δηλαδή, και στη συνέχεια θα απαλωτριώνονται υγιές αυτές. Δεν χρειάζεται να δώσω συγκεκριμένα ονόματα. Ξέρουμε τι παραδείγματα εννοώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος, ο κύριος Αρντός. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στο θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης θα ήθελα να πω το εξή. Έγιναν λοιπόν κάποιες αλλαγές ε, στην Ουγγαρία, στην νομοθεσία σε ό,τι αφορά την ε, πώληση γέων. Ακολουθήσαμε το δανέζικο και γαλλικό μοντέλο, γιατί υποστηρίζω πολύ τις ε, πράξεις διεκτησίας της Δανίας και της Γαλλίας και ως αποτέλεσμα όμως κάποιες χώρες αντιμετωπίσαν διαδικασίες επί παραβάση, οι οποίες ξεκίνησαν εις βάρος τους. Οι Πολωνοί φίλοι μας είναι στην ίδια γραμμή, θα ακολουθήσουν το ίδιο πρόβλημα, θα αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα. Τώρα, για την ελεύθερη κυκλοφορία και το κεφαλαίο. Αυτό απασχολεί τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια σαφή δήλωση ότι τα διπλά μέτρα και σταθμά δεν ε, επιτρέπονται. Το ίδιο που δουλεύει και επιτρέπεται στην Γαλλία και στην Ανία θα πρέπει να επιτρέπεται και στην Ουγγαρία και στην Σλοβακία. Δεν μπορεί να γίνει το διακρίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Πετήρ τώρα. E, Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Νόχιλ για την ε, παρουσίαση που μας έκανε. Να σας πω ότι στην Κροατία πάνω από 90% των ε, οικογενειακών επιχειρήσεων είναι μικρότερα από 9 εκτάρια και ξέρουμε ότι η παραγωγή τροφίμων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ιδιοκτησία των γεωργικών γεών. Άρα θεωρούμε ότι η συγκεντρώση των γεών μέσω μισθώσεων, εκμισθώσεων και καλλιέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν ως ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας. Γιατί μόνο έτσι θα διατηρηθούν οι εταιρείε αυτές. Μόνο έτσι θα συνεχίσουν να επιβιώνουν αυτές οι επιχειρήσεις, να μεταβιβάζουν τις γιες τους νέους, Όλα αυτά εξαρτώνται όμω από τι εθνικέ νομοθεσίε, θεωρώ. Δεν μπορεί να παρέμβει και σε υπερβολικό βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σημείο αυτό. Και αυτό που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει στην Κροατία είναι να οριστεί η βέλτιστη έκταση των γεών βάσει και της περιφερειακής διάστασης της πολιτικής αυτής και θα πρέπει να έχουν δικαίωμα προς υποστήριξη και ενίσχυση οι, οι ιδιοκτήτε. Αλλά θα πρέπει να υποστηρίξουμε γενικότερα τη συγκέντρωση για την εκμετάλλευση και την καλλιέργεια των γεών. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι από την Ανατολική Ευρώπη σε ό,τι αφορά και την εφαρπαγή γεών, του land grabbing, είναι ένα πρόβλημα το οποίο μάλιστα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να γραφτούν κοινέ λύσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Πετήρ. Να πω δύο λόγια πριν δώσω την, ε, το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. σε θέμα, σε θέματα των αρμοδιοτήτων, νομίζω ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ότι αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το θέμα είναι πώ θα βρούμε μια ισορροπία μεταξύ τη υπερβολική ε, συγκέντρωση ή τη ατομική ε, διαμόρφωση ή τη υπερβολική συγκέντρωση. Όταν φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου το 3% των ε, διακριτών έχει 50% των γεών έχουμε πρόβλημα. Αν δεν μπορούμε λοιπόν να παρέμβουμε και να αντιδράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να καταστρέψουμε μια πολιτική για να προωθήσουμε αυτά που επιθυμούμε. Γιατί πλέον ε, έχουμε το φαινόμενο όπου ουσιαστικά η έκταση συνεπάγεται οικονομικό συμφέρον και χρήμα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια βαθμονόμηση, μία εξισορρόπηση της πολιτικής μας για τα επόμενα χρόνια. Αυτό ήθελα να προσθέσω σε αυτή τη συζήτηση. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Βίλμαν. Yes, um, good morning, uh, Καλημέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο που δίνετε το λόγο στην Κομισιόν να παρουσιάσει κάποια στοιχεία στη σημερινή συζήτηση και να εξηγήσει τη δράση της για τη γεωργική γη. Καταρχάς να σας ε, ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι από την ε, Γενική Διεύθυνση ε, Γεωργίας, αλλά ε, σταθερότητα. Λοιπόν, το, το θέμα είναι ε, τι γίνεται με τις ξένες επενδύσεις στην ε, γεωργία και στη γεωργική γη. Να σας εξηγήσω ότι η Κομισιόν πιστεύει ότι συνολικά η ελευθερία επένδυση στην ε, Ευρώπη είναι πολύ θετικό πράγμα. Μπορεί να φέρει σημαντικά πλεονέγματα και στη γεωργική γη και στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Μπορεί, και το έχουμε δει, ε, να φέρει μεταφορά γνώσης, ε, τεχνολογία και να ενισχύσει τη γεωργική παραγωγικότητα. Μπορεί να το κάνει βεβαίως εφόσον υπάρχουν σωστοί κανονισμοί οι οποίοι εξισορροπούν την ελευθερία των επενδυτών με, και την πλαισιώνουν με κανόνες, ούτως ώστε να έχουμε μια βιώσιμη γεωργία και μια σωστή ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση για το νομικό πλαίσιο το οποίο αναφέρα, στο οποίο αναφερθήκατε. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μιλάει ρητά για την πώληση της α, γεωργικής γης. Ε, αλλά όμως δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη ρυθμίζουν αυτό το θέμα. Τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να το κάνουν στο βαθμό που σέβονται τις βασικές αρχές της συνθήκης. Τις βασικές αρχές που είναι οι θεμελιώδες ελευθερίες και κυρίως, και αυτό είναι ο πυρήνας της ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ε, τη μη διάκριση λόγω εθνικότητας. Όταν λέω θεμελιώδεις ελευθερίες, σημαίνει ελευθερία στην κυκλοφορία των κεφαλαίων, και εδώ με αυτό έχουμε να κάνουμε, γιατί η γεωργική γη όντως θεωρείται ως κεφάλαιο και επομένως καλύπτεται από τις συνήθειε διατάξεις της εσωτερικής αγοράς. Και στις ορισμένες περιπτώσεις ε, μπορεί να παίξει ρόλο και η φασική ελευθερία για την ελεύθερη εγκατάσταση. Η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων φυσικά ε, αφορά την εσωτερική ε, αγορά κεφαλαίων και το ίδιο ισχύει για τις επενδύσεις. Και φυσικά ισχύει και για την γεωργική γη. Οι διασυνοριακές επενδύσεις καταρχήν σε γεωργική γη απολαμβάνει τις, ε, των τεσσάρων ελευθεριών. Δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός για κάτι τέτοιο. Αυτό το λέει το άρθρο 63 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι ξεκάθαρο και από τις άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Όμως νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι υπάρχουν ατότητες περιορισμών σε αυτές τις ελευθερίες όταν είναι απαραίτητες για να υπερασπίσουν και να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον. Εμείς πιστεύουμε ε, ότι οι συνθήκες αφήνουν τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ακούστηκαν στη σημερινή συζήτηση. Πιστεύουμε ότι επειδή υπάρχει επαρκής νομολογία για την αγορά γεωργικής γης, ε, η οποία επιβεβαιώνει ότι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνώρισε την ιδιαίτερη φύση της γης και την ανάγκη να την προστατεύσουμε. Έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας για να την προστατεύσουμε λοιπόν. Λοιπόν, θα δώσω κάποια παραδείγματα. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων μπορεί να περιοριστεί για να εμποδίσουμε την κερδοσκοπία γης. Το δικαστήριο είπε ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να Ε, κρατήσουν ε, παραδοσιακές μορφές ε, καλλιέργειας όπως την οικογενειακή γεωργία. Συμφωνεί επίσης ε, με την αρχή ότι η γεωργική γη πρέπει να πηγαίνει καταρχήν στους γεωργούς. Επομένως όλα, τα, όλα αυτά τα, θέματα που είναι θέματα δημοσίου συμφέροντος μπορούν να δικαιολογήσουν την, τον περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία. Μπορούν να δικαιολογήσουν και το τονίσω. Γιατί οποιοδήποτε περιορισμός, και πρέπει να το πούμε εδώ, θα πρέπει να δικαιολογείται. Μόνο όταν υπάρχει δηλαδή δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή οι περιορισμοί θα πρέπει να είναι αναλογικοί για να είναι αιτιολογημένοι. Δηλαδή δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν το απολύτως απαραίτητο για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος. Αυτά ήθελα να πω. Να σας πω δηλαδή ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει ειδική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα κράτη-μέλη έχουν τους νόμους και ρυθμίζουν κτλ. Και, και πρέπει να σέβονται απλώς τις βασικές αρχές της συνθήκης που παράλληλα επιτρέπει να πάρουμε προστατευτικά μέτρα ε, για να περιορίσουμε τους κινδύνους για το δημόσιο συμφέρον. Αυτό το πλαίσιο έπρεπε να το πούμε, γιατί ακούστηκαν τόσες ανησυχίες για τις ξένες επενδύσεις. Οι ξένες επενδύσεις σε γεωργική γη ε, στην πραγματικότητα είναι πολύ περιορισμένοι. Δεν είναι εύκολο να έχει κανείς αξιόπιστα, αξιόπιστα στοιχεία, αλλά από τις πληροφορίες κομισιών το ποσοστό των γεωργικών γεών που ελέγχουν οι ξένοι επενδυτές κτλ. είναι πολύ χαμηλό. 1 με 3% με βάση πληροφορίες που έχουμε. του λεχθέντος σημειώνουμε ότι υπάρχουν εκθέσεις, ότι οι ξένες επενδύσεις αυξάνονται και ότι υπάρχει ολένα και μεγαλύτερη όρεξη για αγορά γης τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά θα πρέπει να προσέξουμε τέτοιο φαινόμενο. Να σας ενημερώσω πριν κλείσω για τη νομική δράση της ε, Κομισιόν ε, πρόσφατα για τον καονισμό για τη γεωργική γη. Αν ξέρετε, το 2014 και 2016 ε, τέλειωσαν οι μεταβατικές περίοδοι μέχρι των οποίων τα κράτη-μέλη τα οποία μπήκαν το 2004 και 2007 θα μπορούσαν να παρεκκλίνουν από τις αρχές των, της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων. Επομένως, αυτές οι χώρες για κάποιο χρονικό διάστημα ε, μπορούσαν να περιορίσουν την αγορά γεωργικής γης από τους ξένους για το χρονικό διάστημα που θεωρούσαν, θεωρούσαμε απαραίτητο για να προετοιμαστούν οι αγορές ε, γεωργικών γεών για μια πιο ε, ελεύθερη αγορά. Έκτοτε, διάφορες χώρες υιοθέτησαν νέους νόμους για να ρυθμίζουν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Έχουμε λάβει τεράστιο αριθμό παραπώνων εναντίον αυτών των νόμων και χρειάστηκε να αντιδράσουμε. Τελικά, κάποιε από αυτέ τι εθνικέ ρυθμίσει τι αμφισβητήσαμε και προσφύγαμε εναντίον, γιατί κατά τη γνώμη μα παραβιάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων κυρίω. Οι διαδικασίε ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2015 και μέχρι στιγμή αφορούν τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, αλλά όχι τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Έτσι. Στη Ρουμανία δεν ε, βρήκαμε να υπάρχει πρόβλημα στην νομοθεσία της. Το Μάιο του 2016 η Κομισιόν πέρασε στην επόμενη φάση διαδικασίας που είναι η τελευταία φάση. Ε, πήγαμε στην αιτιολογημένη έκθεση δηλαδή ε, πριν πάμε στο δικαστήριο. Μέχρι στιγμής εξετάζουμε τις απαντήσεις στις επιστολές που στείλαμε δεν ξέρω τι θα γίνει στην επόμενη φάση, αν θα πάμε τελικά, αν θα προσφύγουμε στο δικαστήριο εναντίον των χωρών αυτών, γιατί ενημερωθήκαμε ότι διάφορες χώρες έχουν ε, ή ετοιμάζουν νομοθεσία για να ε, αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και θα πρέπει να εξετάσουμε αυτή τη νέα νομοθεσία. Αλλά μπορώ να σας ε, κάνω μια σύντομη επισκόπηση κάποιων από τα προβλήματα που εντοπίσαμε. Η βασική ανησυχία στη Βουλγαρία και στην Σλοβακία είναι ότι οι, αγορε... οι αγοραστές θα πρέπει να είναι μακρά διαμένοντες στις χώρες αυτές ε, που νομίζω ότι είναι μια διάκριση βάρων άλλων Ευρωπαίων υπηκών, η Ουγγαρία. Είναι, ε, έχει ένα σύστημα πολύ περιοριστικό, με πάρα πολλές προϋποθέσεις για την αγοραγής. Μεταξύ άλλων, υπάρχει ε, πλήρης απαγόρευση αγοράς γεών από, φυσικά, από νομικά πρόσωπα, το οποίο ε, εμείς το αμφισβητούμε. Και επίσης στην Ουγγαρία και στη Λιθουανία θα πρέπει να είσαι αγρότης για να μπορέσεις να αγοράσεις αγροτική γη. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις έχουν εισαχθεί υποτίθεται για το δημόσιο συμφέρον, για να μειωθεί η κερδοσκοπία και να διατηρηθεί η χρήση της ε, γεωργικής γης για γεωργικούς λόγους. Η Κομισιόν δεν αμφισβητεί ότι αυτοί οι στόχοι είναι θεμητοί, ότι είναι καλοί, ότι πρέπει να υλοποιηθούν. Απλώς κάποια από τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί δεν είναι αναλογικά, υπό την έννοια ότι κάποια άλλα λιγότερο περιοριστικά μέτρα θα μπορούσαν να εξίσου αποτελεσματικά για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Κάποια από τα μέτρα επίσης ε, εισάγουν ε, διακρίσεις, όχι άμεσα, αλλά de facto για λόγους εθνικότητας. Ε, Δηλαδή, το γεγονός ότι ο αγοραστής θα πρέπει να διαμένει στη χώρα ή και στο Δήμο μάλιστα, για, ε, στον οποίο ανήκει η γη για να μπορέσει να τα αγοράσει, είναι τεράστιος περιορισμός. Προκύπτει από την νομοθεσία ότι αυτή η ρύθμιση παραβιάζει την ενωσιακή νομοθεσία. Και άλλη μία ε, νομική λεπτομέρεια. Ε, γιατί είπατε εσείς ότι η γη πρέπει να αγοράσετε από τους γεωργούς. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι οι πωλήσει ε, μπορεί να υπόκεινται σε πρώτερη έγκριση από τις δημόσιες αρχές. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να εξασφαλίσει ότι υπό κάποιες συνθήκες οι γεωργοί έχουν την προτεραιότητα να αγοράσουν τη γεωργική γη, δηλαδή προτεραιότητα έναντι άλλων, ε, μέσω δικαιωμάτων προαγοράς φερρυπίν. Ε, επιτρέπ, αυτά ήταν κάποια συμπεράσματα. Τώρα, κάποια συμπεράσματα. Ε, οι σε επιβαραβάση είναι σε φάση εξέλιξης ε, για τα κράτη-μέλη που σας ανέφερα και ελπίζουμε τελικά να βρούμε λύσεις οι οποίες ε, αντιμετωπίζουν επαρκώ τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε ε, και παράλληλα ε, χωρί να παραβιάζουμε και την ενωσιακή νομοθεσία. Επίσης, η δράση αυτή ευθυγραμμίζεται μετά όσο έχει κάνει η Κομισιόν στο παρελθόν σε σχέση με τους καονισμούς. Στο παρελθόν τα τελευταία δέκα χρόνια η Κομισιόν έχει προβεί σε διάφορες ε, δράσεις. Ε, έχουμε δηλαδή επαρκή νομοθεσία του, νομολογία συγγνώμη, του δικαστηρίου για όλα αυτά τα θέματα και η Κομισιόν τέλος θα λαμβάνει συνέχεια ε, πληροφορίες για το δίκαιο περί διοκτησίας από όλα τα κράτη-μέλη. Συχνά λαμβάνουμε πληροφορίες μέσω παραπώνων που υποβάλλουν ε, οι πολίτες. Ε, παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Είμαστε οι θεματοφύλακες των συνδικών και είναι το καθήκον της Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι το δίκαιο γίνεται σεβαστό και να λάβει νομική δράση εάν χρειάζεται. Ε, πολλές ε, φορές ακούσατε, ακούσαμε να μιλάτε για κατευθυντήριες γραμμές. Ε, και ζητάτε να υπάρξουν κατευθυντήριε γραμμέ ε, στην Ένωση. Τέλο πάντων, περιμένουμε λοιπόν ε, την έκθεσή σα για να μπορέσουμε να τη διαβάσουμε. Ευχαριστούμε. Κυρία Νόιχλη, για δύο λεπτά. Ούτε καν δύο λεπτά χρειάζομαι. Δύο φράσεις μόνο. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά σας. Ε, θα τα γράψω, τα σημείωσα και όλα αυτά. Ενδεχομένω να σα ρωτήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω το εξή. Το χθε ήταν χθε, το παρελθόν. Σήμερα έχει αλλάξει η αγορά. Είναι διαφορετική η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσαρμοστεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις ε, πρέπει να πω ότι λυπάμαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά μόνο αντιδράει στα σχόλια των ε, κρατών μελών με επιστολές, με θυμωμένες επιστολές, αντί να δρά ενεργά για την προστασία των ε, καλλιεργήσιμων γεών. Αυτό είναι και θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το πώς μπορούν να προσαρμοστούν πώς μπορούν να προστατευθούν τα συμφέροντα των κρατών μελών και να αποφασίσει με τον ε, στόλο, με τον μεγάλο στρατό των δικηγόρων που έχει, τι εργαλεία επιτρέπονται. Το θέμα της ισορροπίας σε ό,τι αφορά την διεκτησία έχει να κάνει με την ε, διατήρηση κάποιων λεπτών ισορροπιών στον κοινωνικό ιστό. Και θα πρέπει λοιπόν πάντα να έχουμε υπόψη ότι το θέμα της ιδιοκτησίας γεών είναι σημαντικό. Και σε αυτό το συγκείμενο λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε την έκθεση αυτή, γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την επιθυμία των κρατών μελών να προστατεύουν τις γέες τους και προβλέπω στη μελλοντική συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Μαρία, σας ευχαριστούμε για αυτές τις διευκρινήσεις. Ε, αυτό το... Ε, στις 10 Νοεμβρίου θα εξετάσουμε την έκθεση. Ευχαριστούμε. Θα δώσω τον λόγο στον πρόεδρό μας για να συνεχίσουμε τις εργασίες. Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας, κύριε Ντάντα. Το πρόβλημα της συγκέντρωσης γεών, ναι, είναι και πρόβλημα αποτελεσματικότητας, ε, ανταγωνισμού. Πρόκειται για σημαντικά πολιτικά προβλήματα, μίλησε εξάλλου για αυτά και ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φυσικά, ε, Θέλουμε να υπερασπιστούμε τη γεωργία, αλλά υπάρχουν και παράμετροι που δεν σχετίζονται με τη γεωργία. Φυσικά, είναι θέμα ε, προσόδων, ε, θέσεων εργασίας, ανταγωνιστικότητας. Ε, υπάρχουν διάφορες διαστάσεις που πρέπει να συμπολογίσουμε διότι σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της παραγωγής. Μειώνεται η παραγωγικότητα, μειώνονται οι πρόσοδοι, μειώνεται η ανταγωνιστικότητά μας σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Και μην ξεχνούμε ότι το θέμα συνδέεται με την οικονομική κατάσταση. Στα νέα κράτη-μέλη υπάρχουν κάποιοι de facto περιορισμοί Η Γεωργή στα νέα ε, δεν είναι κατά της ε, μεταπόλησης ε, των γεών, στο μέτρο όμως που είτε θα συνεκμεταλλευτούν ε, το αγροτεμάχιο είτε θα το εκμεταλλευτούν οι ίδιοι. Και δεν μιλάμε μόνο για ε, επενδύσεις μεγάλου κεφαλαίου, αλλά υπάρχουν και αυτά τα κινήματα των γεωργών. Λοιπόν, πρέπει να εξετάσουμε το θέμα από πολιτικής πλευράς, από οικονομικής πλευράς και να μην ξεχνούμε το θέμα της πρόσβασης ε, στη γη. Μία, όταν ένας γεωργός ή μια γεωργική εκμετάλλευση θέλει να αγοράσει γη, αυτό φέρνει έσοδα, φέρνει Ε, και πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Λοιπόν, ε, ας περάσουμε στο επόμενο σημείο ε, της ημερήσιας διάταξης. Θα ανταλλαγεί απόψε με έναν εκπρόσωπο του Παγκοσμίου Φόρουμ για την πρόσβαση στους φυσικούς πόρους στην Βαλένθια, στην Ισπανία, έγινε η τελευταία συνεδρίαση αυτού του φόρουμ. Ε, στον τον Απρίλιο του 2016 πάνω από 1.200 οργανώσεις, εθνικές οργανώσεις, ενώσεις γεωργών, ε, οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών, διεθνείς και εθνικές οργανώσεις από 70 χώρες 400 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτή την ανοιχτή συζήτηση σε σχέση με την πρόσβαση στους φυσικούς πόρους. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μισελ Μεχλέ από την οργάνωση ΑΚΤΕΡ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σας δίνω λοιπόν μέσω το λόγο. Η οργάνωσή σας ναι, έχει πολύ σημαντικό ρόλο για το θέμα της πρόσβασης των φυσικών πόρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είναι μεγάλη τιμή για μένα να μπορέσω να σας παρουσιάσω τη, τα αποτελέσματα αυτού του, των εργασιών αυτού του φόρουμου. Ευχαριστούμε, κύριε Νόχη που προτείνατε να παρέμβουμε στα πλαίσια της σημερινής συζήτησης. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πολύ πιο εντατικά συμμετείχαν στη διοργάνωση αυτού του φόρουμ. Ο, ο κύριος Τσιάλος ε, συνδέχτηκε η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Άγκρη να είναι μία από τις οργανώσεις που ζητούν τη διοργάνωση του φόρουμ. Δυστυχώς όμως με την αλλαγή του Επιτρόπου Λίγο πριν αποχωρήσει από θέση του ο κ. Στάσιαν ε, μαζί της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποχωρήσει από τις οργανώσεις που ζητούσαν τη ε, διοργάνωση του φόρουμ. Έγιναν πολλέ συνεδριάσεις, ποτέ δεν αποκαταστάθηκε ο διάλογο. Θα μα επέτρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετέχει σε αυτή την διοργάνωση. Είναι κρίμα. Αντίθετα, ε, είχαμε την υποστήριξη της ΕΟΚΕ ε, και κάναμε και μία προπαρασκευαστική. Συνεδρία στα τέλη του 2015 θα επανέλθω σε αυτό και συμμετείχαν και διάφοροι ε, βουλευτές ε, που εκπροσωπούσαν ε, τις δικές τους οργανώσεις, εθνικές οργανώσεις. Ε, λοιπόν, ε, δέκα χρόνια μετά, μετά την παγκόσμια διάσκεψη του ΦΑΟ στο Πόρτο Αλέγκρι το 2016 για την πρόσβαση στη γη και τους φυσικούς πόρους, βλέπουμε ότι το θέμα της, ε, του ιδιοκτησικού καθεστώτος είχε αναπτυχθεί με τρόπο αντίθετο από αυτό που ζητούσε λοιπόν το φόρουμ στο Πόρτο Αλέγκρε. Ε, σε παγκόσμιο επίπεδο είχε επιδεινωθεί τόσο η κατάσταση που σε παγκόσμιο επίπεδο θα έπρεπε να διοργανώσουμε ένα φόρμα να συμμετέχουν οι κυβερνήσει, οργανώσει κοινωνία των πολιτών αλλά και ειδικοί εμπειρογνώμονε οργανώσει που γύθηκαν τη διαδικασία ε, το Σεράγι, μια μικρή ισπανική οργάνωση και η ΆΚΤΕΡ, η δική μας οργάνωση, πολύ γρήγορα ε, βρήκαν πολύ άριθμε οργανώσεις που υποστήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και δεν θέλω να σα το κρύψω, είχαμε πελώρες δυσκολίε. Ε, καταφέραν παρόλα αυτά από 70 χωρί για τρει ημέρε να έχουμε 400 ανθρώπους από καπαόμικρον βοσκούς, γεωργούς, και με εκπροσώπους όμως και των κυβερνήσεων από το Υπουργείο Γεωργίας Γαλλίας και διάφοροι ακαδημαϊκοί. Ε, υπάρχει μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα που ε, υπάρχουν τα στοιχεία για την διοργάνωση του φόρουμ. Ε, θα επικεντρωθώ σε σημαντικά συμπεράσματα. Θέλαμε να κάνουμε με προπαρασκευαστική συνεδρίαση αναήπειρο στην Ευρώπη. Κάναμε την επίσημη συνεδρίαση σε συνεργασία με το, ε, την ΕΟΚΕ, όπως σας είπα. Εκεί διαπιστώσαμε ότι ε, ε μεταρρυθμίζεται ε, άρδιν η γεωργική παραγωγή, μεγάλη πόλη, μεγάλη συγκέντρωση των γεών πέρα από την υφαρπαγή με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Ε, πρόκειται για βαθιά ριζική αλλαγή του γεωργικού κόσμου στην Ευρώπη που και πάλι δημιουργεί το δίλημα ποιο μοντέλο γεωργικό θα πρέπει να επιλεγεί. Είναι μια ε, επιλογή και κοινωνικού χαρακτήρα και πρέπει να γίνει. Αυτό έγινε εξάλλου δεκαετία του 60 στις αρχές της κοινή γεωργικής πολιτικής όμως ε, είναι πλέον απαρχαιωμένες αυτές οι αποφάσεις ε, και δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση με αυτά που επιθυμούσαν οι ιδρυτές της το 60. Ε, βλέπετε τα πρακτικά από τη συνεδρίαση που κάναμε. Donc, vous trouverez le compte rendu de cette réunion. Πρακτικά τη συνεδρίαση του Νοεμβρίου για, ε, βρίσκεται στη, στο, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα επανέλθω σε κάποια στοιχεία κατά τη διάρκεια της παρουσίασής μου. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα του Παγκοσμίου Φόρουμ για την πρόσβαση στη γη ότι είναι εφαρμόσιμα ε, σε παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτά τα πορίσματα. Το πρώτο πράγμα από το οποίο καταλήξαμε σε συνένεση είναι ότι μεταξύ των μεγαλύτερων παγκοσμίων προκλήσεων υπάρχει σοβαρή αντίφαση ανάμεσα στον καπιταλιστικό κόσμο των μισθωτών και το, τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Σε κοινωνικό επίπεδο εκφράζεται αυτή η διαφορά γιατί υπάρχει το θέμα της απασχόλησης. Σε οικονομικό επίπεδο σε σχέση με την προστιθέμενη αξία ανά εκτάριο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο διατήρησης βιοποικιλότητας, ε, της παραγωγικότητας ε, των εδαφών, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Ε, όλοι οι μετέχοντες στο φόρουμ, ανεξαρτήτως προέλευσης, συμφώνησαν ότι η παραγωγή ε, από πλευρά των γεωργών ή ε, οικογενειακών εκμεταλλεύσεων ως προς την προσθέμενη αξία ανακάτοικο είναι πολύ υποφελέστερη για το σύνολο του κοινωνικού ιστού σε σχέση με την μεγάλη βιομηχανική γεωργική παραγωγή. Αυτό είναι γενικότερο συμπέρασμα και είπε εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρόκειται για την εξυπηρέτηση του κοινού ενδιαφέροντο. Ναι, περί αυτού πρόκειται. Ποιε μορφέ γεωργική παραγωγή μα επιτρέπουν λοιπόν να εξυπηρετήσουμε το κοινό γενικό καλό η συγκέντρωση των πόρων και των γεών σε λίγα χέρια, σε λίγους ιδιοκτήτες με ε, συγκέντρωση αλλά και η φαρπαγή παραβίαση των δικαιωμάτων των πιο πληθυσμών ε, συνιστά ε, μία παραβίαση των δικαιωμάτων γενικότερο πέρα από αυτούς τους ανθρώπους που πλήττονται άμεσα ε, αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε, διότι εάν εστιάζουμε σε αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το θέμα της υφαρπαγής, ε, παραγνωρίζουμε τη σημασία των οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ε, τρίτο βασικό συμπέρασμα, η απελευθέρωση των ανταλλαγών των γεωρικών αγαθών σε παγκόσμιο επίπεδο και ταυτόχρονα υποστήριξη των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι οι δύο βασικές αιτίε αυτή τη δυσμένου εξέλιξη. και ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αύξηση ανταγωνιστικότητας ανάμεσα σε γεωργούς ε, των οποίων η παραγωγικότητα παρουσιάζει μεγάλε διαφορέ και πλήττονται οι λιγότερο παραγωγικοί φυσικά συστηματικά ω προ το κόστος εργασία να το τονίσουμε αυτό, πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στην παραγωγικότητα συνεργασία σε σχέση με την παραγωγικότητα καθαρού πλούτου ανά εκτάριο, διότι αυτοί που έχουν την υψηλότερη παραγωγικότητα προς το εργασιακό κόστος, ποιοι είναι αυτοί που έχουν λίγους μισθωτού ε, ανά εκτάριο, όμως ανά εκτάριο ταυτόχρονα παράγουν τη μικρότερη προστιθέμενη αξία. Ε, το μικρότερο καθαρό πλούτο, οπότε αυτό είναι, δεν είναι υποφελέ για την κοινωνία, διότι πλήττονται οι φτωχότεροι σε αυτή την περίπτωση και με τις παρεκβολές που μπορέσαμε να κάνουμε εκτιμήσαμε ότι αν σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμόζουμε την πολιτική που εφήρμοσε η Γαλλία στη δεκαετία του 60 ή και νωρίτερα και μέχρι σήμερα δηλαδή εάν μειώναμε τον ενεργό γεωργικό πληθυσμό σε 2-3% σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι το 2005 για να έχουμε πλήρη απασχόληση θα έπρεπε ε, να φτιάξουμε νέες θέσεις εργασίας. 3-4 δισεκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Αδύνατο. Μπορούμε να κάνουμε για τον υπολογισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την υποαπασχόληση και την ανεργία. Δεν έχει νόημα όμως ε, σήμερα να δημιουργούμε εξαιρετικά αποτελεσματικές ε, γεωργικές επιχειρήσεις που όμως δεν έχουν υπαλλήλου, δεν έχουν μισθωτούς ε, και ξαναλέω έχουν πολύ μικρή προσθέμενη αξία ανά ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά ενετικές επιπτώσεις ε, για την περιβαλλοντική διάσταση. Πολύ βασικό συμπέρασμα του φόρουμ, λοιπόν, το θέμα, τα οικονομικά ζητήματα και τα θέματα του, ε, των της κοινοφελούς υπηρεσίας πρέπει να μπουν στον πυρήνα της όλης της διαδικασίας. Ε, πάνω από 50% του πληθυσμού της γης ε, είναι, ζουν στην Ήπεθρο και δεν μπορούμε πλέον να... Ε, ε, ξεχνούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές και άρα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αναθεώρηση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Ε, δεν μπορούμε να πείσουμε λοιπόν Αλλιώ ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τις ε, μελλοντικέ εργασίες οι, αστι... οι οργανώσεις που χειρίζονται το αστικό περιβάλλον ή και το περιαστικό περιβάλλον δεν μπορούν να μην ασχολούνται με την αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής γιατί του αφορά. Αυτό πρέπει να αλλάξει πλέον και αυτό, σε αυτό το συμπέρασμα καταλήξαμε στο Παγκόσμιο Φόρουμ. υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που είπαμε. Τα πρακτικά ακόμη τώρα τα ετοιμάζουμε. Δεν σε επεκτάθω. Επανέρχομαι στην Ευρώπη. Ε, απαρίθμησα τώρα όλα τα έγγραφα που χρησιμοποίησαμε ως βάση των συζητήσεων. Δεν βλέπετε όμως τίποτα γιατί ε, ε, αυτό είναι χαρακτηριστικό ενός κακοφτιαγμένου PowerPoint, γιατί είναι πνιγμένο στο κείμενο και δεν μπορείτε να διαβάσετε τίποτα. Αν θα, σας δώσουμε θα σας δώσουμε όλους τους συνδέσμους. Ε, υπάρχει μια μελέτη της Via Campesina Ευρώπη, ή το μελέτη του ΣΕΖ, ε, του, της ΕΟΚΕ δηλαδή, μελέτη που ζήτησε το Κοινοβούλιο από το Ινστιτούτο Τρανσνάζ και μελέτες που έγιναν από οργανώσεις όπως σας αφέρει στη Γαλλία ή οργανώσεις που ασχολούνται με την ε, δομή, με το ειδικτυσιακό καθεστώς των γεών στην Ευρώπη. Δεν είναι θέμα δεξιάς και αριστεράς, είναι θέμα επιλογής του κοινωνικού μοντέλου για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δυστυχώ ε, δεν, ε, επειδή έφτασα λίγο αεροπορημένο, ε, γιατί είχα το τραμ. Τι να κάνω, συμβαίνουν και αυτά στο, στα πράστια, στο Παρίσι και έχασα τη μισή παρουσίαση της κυρίας Νόξιλ, αλλά άκουσα διάφορες παρατηρήσεις που ε, εντάσσονται σε αυτά που σας είπα και εγώ για την ιστορία του για τους στην Ευρώπη. Ε, επίσης, μην ξεχνάμε ότι οικοδομήσαμε την ανάπτυξη συνειδητά επί τη βάση της γεωργικής παραγωγής εδώ στην Ευρώπη. Επί τη βάση των ε, ε, γεωργικών, ε, των οικογενειακών εκμεταλλευτών. Όχι παντού, όχι με ομοιόμορφο τρόπο, αλλά δεν επικρατούσαν τα Ποια είναι η ΚΑΠΑ. Ο στοχο είναι η αυτάρκεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επαρκή εισοδήματα για του παραγωγού και όχι για του ιδιοκτήτες, όχι για το κεφάλαιο. Είναι Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση και ε, τιμές προσιτές δικές από τους καταναλωτές, αλλά και εξυγχρονισμός Τη γεωργίας και εξαγωγές των προϊόντων. Ε, η κατάσταση στα κράτη είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με πριν από μία πενταετία και παρουσιάζει μεγάλες διακοιμάνσεις σήμερα. Ε, είναι, θα έλεγα, διαπιστώνουμε ξενόμενη πόλωση και συγκέντρωση των γεών μεγάλε καπιταλιστικέ ε, καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις ε, με μισθωτούς που προέρχονται από το κληροδότημα της ε, καταναγκαστικής κολεκτιβοποίησης των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης με αποκατάσταση του δικτυσιακού καθεστώτος που όμως δεν εμπόδια τη συγκέντρωση ε, σε αυτέ τι μεγάλε εκμεταλλεύσει. Ε, μην ξεχνάμε, οι εκμεταλλεύσει είναι μισθωτέ ε, και όχι ιδιοκτήτε, όπω στη Ρουμανία το άκουσα, το είπατε. Και σε αυτέ τι χώρε τη παλιά Ευρώπη. Ε, τώρα δεν είναι πολύ εύστοχο να εκφράζουμε έτσι, αλλά ήθιστε. Στη Γαλλία, παραδείγματο χάρη, βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο ένα και περισσότερες εταιρείε ε, γεωργοί που διαχειρίζονται τα γεωτεμάχια με ε, συλλογικό τρόπο ε, και επηρεάζεται ο τρόπος λειτουργίας, δηλαδή βλέπουμε τον μικρό γεωργό που προσπαθεί να διατηρήσει το κληροδότημα για τις επόμενες γενιές λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές ε, ανάγκες και όλα αυτά υποχωρούν διότι σκεφτόμαστε, σκέφτονται οι μεγάλες εταιρείες ως μέτοχοι παρότι σε, οι μέτοχοι είναι μέλη οικογενειών. Αλλάζει όμως η λογική και δυσκολεύεται, δυσχεραίνεται ε, η ρύθμιση της ε, αγοράς για την πρόσβαση στις αγοραπολισίες των γεωτεμαχίων. Έχουμε την εκμίσθωση με το νέο νομοσχέδιο και δεν ρυθμίσαμε τα κοινωνικά μερίδια. Δηλαδή, ε, μπορεί ε, εκατομμύρια εκτέρια να αγοράζουν κινέζικες εταιρείες ε, ή παίρνουν ταμπέλια χωρίς να υπάρχει κανένας μηχανισμός ελεγκτικός ταυτόχρονα. Πλήρης είναι η σύγχυση ελεγκτικος ταυτοχρονα πλήρη ειναι η συγχυση αναμεσα σε αυτούς που υπερασπίζουν τη λογική των μικρών γεωρικών μεταλλεύσεων και αντίθεσή του αυτούς που στηρίζουν τη λογική των μεγάλων γεωρικών εταιρείων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 συνεχίσουμε τη συζήτηση θα πρέπει να μην ενδιαφερόμαστε μόνο στο θέμα της κατανομής ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά και στο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπορούμε να αφήσουμε την ιδιοκτησία χωρίς να την αλλάξουμε και ε, να ρυθμίζουμε το μέγεθος, ε, δηλαδή τι μπορεί κάποιος να παράξει. Δεν έχει σχέση ε, το δικαίωμα παραγωγής με το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Η εκμίσθωση είναι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη ε, έγινε η ανακατανομή τη ιδιοκτησία στη Ρουμανία παραδείγματο χάρη και στην Ουκρανία έτσι μετά την αποκολεκτιβοποίηση δεν του αφήσαμε όμω, αυτοί που πήραν αυτά τα μικρά αγροτεμάχια Πώ να τη μετατρέψουν σε γεωργικό τεμάχιο, σε ε, ε, ε, οικογενειακή εκμετάλλευση. Ε, ανοίξαμε τα παραθυράκια λοιπόν στο μεγάλο κεφάλαιο για να φτιάξουν μεγάλε μεγάλες εκμεταλλεύσεις. δεν τα έχω κατά ξέρετε τα νούμερα, τα ίδια, ξέρετε καλύτερα από μένα στη Ρουμανία. Ε, πάνω από 50.000 εκτάρια, μία εκμετάλλευση στη Ρουμανία. Κάντε μία σύγκριση με το μέσο όρο τη Γαλλία, 60 εκτάρια ή με την κατάσταση είπατε 10 εκτάρια σε άλλες χώρες, καταλαβαίνετε ότι έχουμε βραζιλοποιηθεί, δηλαδή ο μεξικοποιηθεί, ε, όπως ήταν η κατάσταση στις αρχές του 20ου αιώνα, εξε, ακραία πόλωση και αυτό οδήγησε στην επανάσταση στο Μεξικό. Ε, κοινωνικές αναταραχές ε, μπορεί να πάρει διαφορετική μορφή αντίδραση εδώ, αλλά αυτή η πόλωση, η φαινόμενη πόλωση, δημιουργεί πρόβλημα διότι δεν έχουμε την κατάσταση πλήρους απασχόλησης δεκαετία του 60, όπως ήταν στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης όταν ξεκίνησε η, η γεωργική πολιτική. Λοιπόν, η ύπεθρο και το αστικό περιβάλλον πρέπει να συνδυαστούν και έχουμε νέου περιβαλλοντικού περιορισμού και το θέμα των εσωτερικών και εξωτερικών μεταναστεύσεων. Πώ όλα αυτά συνδέονται με την βελτιστοποίηση τη χρήση τη υπαίθρου. Επαναπροσδιορισμό λοιπόν της γεωργίας ε, σε σχέση με αυτά που χρειαζόμαστε αρχές του 20ου αιώνα και φυσικά αυτό πρέπει να γίνει διαφορετικά σε κάθε κράτος μέλος, όμως ταυτόχρονα πρέπει να κινηθούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να αφήσουμε την Ευρώπη να προωθεί την απελευθέρωση των κεφαλαίων, εάν ναι, αυτή η απελευθέρωση των κεφαλαίων ναι, θέτει να αμφίβολο την πολιτική, όπως ακούσαμε και στη δική σας συζήτηση, της ε, στήριξης προς την οικογενειακή γεωργία που υπάρχει σε, κάποια, ε, σε κάποιες χώρες για την συμμετοχή στο Παγκόσμιο φόρμα για την πρόσβαση στη ε, βασιζόμαστε στην οικογενειακή γεωργική παραγωγή σε εθνικό επίπεδο που σχετίζεται με τι γειτονικέ αστικέ περιοχέ. Μόνο έτσι μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε το γεωργικό μοντέλο και αυτό. Συνεπάγεται εξουδετερώση σημαντικών λόμπι που όπω ξέρουμε επηρεάζουν ε, πάρα πολύ τι αποφάσει που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. En fait, il y Λοιπόν, τώρα ε, χοντροειδώς, δύο προτάσεις. Θα πρέπει να σταματήσουμε την ε, πόλωση αυτή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και θα πρέπει να ε, διευκολύνουμε την εγκατάσταση νέων γεωργών. Αυτό ισχύει παντού. Και στην Γαλλία και στη Ρουμανία, στην Αγγλία, οπουδήποτε. Παντού. Δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουμε την ε, αγροτική γεωργική λογική με την ε, λογική των, ε, της μετοχικής εταιρεία. Θα πρέπει να κρατήσουμε την αρχική λογική ας πούμε, της οικογενειακής παραγωγής στη γεωργική και να μην περάσουμε στη λογική του κεφαλαίου. Γιατί αν περάσουμε στη λογική της μεγιστοποίησης ας πούμε, των επενδύσεων και του μέγιστου κέρδους, στην πραγματικότητα θα προωθήσουμε φιλελεύθερη, μια ε, φιλελεύθερη, ακραία φιλελεύθερη ας πούμε, πολιτική στη Γεωργία ε, εις βάρος του συνόλου του ε, ευρωπαϊκού πληθυσμού. Θέλω να κάνω δύο μεγάλες, δύο αδρές προτάσεις, που είναι ιδέες, τις οποίες πρέπει να εξετάσουμε λιγάκι. Δεν τα ξέρω όλα αυτά λεπτομερώς. Τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Νομίζω ότι θα πρέπει να τροποποιήσουμε τις πολιτικές και τα εργαλεία της Ευρώπης. Όταν αυτά τα εργαλεία ε, επιτείνουν μια, κάποιες καταστάσεις που είναι αντίθετες προς το συμφέρον της Ευρώπης. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Σημαίνει διάφορα πράγματα. Σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναδούμε την ε, ε, κατανομή των ενισχύσεων της κάτω. Όταν κάναμε αυτή την ε, συνεδρίαση τον Νοέμβριο του 2015 είχαμε πει ανώτατα όρια στις επιδοτήσεις. Επίσης αντί να επιδοτούμε ε, αναεκτάριο, να δίνουμε τις ενισχύσεις δηλαδή εκτάριο, Παραδείγματο χάρη, αν έχουμε 10.000 εκτάρια, παίρνουμε 10.000 φορέ περισσότερη βοήθεια από αυτόν που έχει ένα εκτάριο, να ενισχύουμε αυτού που είναι ενεργοί. Επίση, αντί να βοηθάμε την παραγωγή αγροκαυσίμων, θα πρέπει να παράγουμε τρόφιμα και επίσης ενίσχυση για το σεβασμό του περιβάλλοντος. Όλα αυτά μπήκαν ε, εν μέρη στην τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, αλλά όχι πλήρω υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν ακόμα. Και θα πρέπει να αφήσουμε μεγαλύτερη ελευθερία στις χώρες ώστε να έχουμε προσαρμοσμένε πολιτικέ στη δική του πραγματικότητα και επίση, τελειώνω, να αυξήσουμε τις βοήθειες ε, προς τις χώρες ε, για να μπορέσουν να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος. Ειδικά στις νέες χώρες γινόταν παλιά, τώρα δεν γίνεται. Επίσης, να περιορίσουμε στην έγκυα ιδιοκτησία αυτή την ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου, ξεκινώντας από αυτή την παλιά διαπίστωση οικονομικής φύσεως, ότι δηλαδή η γη δεν είναι κεφάλαιο όπως οτιδήποτε άλλο. Το να θεωρήσουμε ότι η γη είναι κεφάλαιο όπως ένα άλλο αγαθό, ας πούμε, είναι ε, η απαρχή όλων των λαθών που είδαμε. Και δεύτερον, για να μην ε, ξεπεράσω πολύ το χρόνο μου, να διευκολύνουμε σε επίπεδο κάθε κράτους μέλους ε, πολιτικές ε, ρύθμισης της ε, έγκυας αγοράς, της έγκυας ιδιοκτησίας, αγοράς και μίστοσης ε, και της, την αγορά, την προώθηση μιας γεωργίας η οποία να εδράζεται στο, στην περιοχή, ας πούμε, στην Ήπεθρο, στο περιβάλλον αυτό, με την επιστροφή στη γη κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είναι περιθωριοποιημένοι οικονομικά και που είναι όμως, οικονομικά είναι ασήμαντοι λοιπόν, αλλά κοινωνικά είναι σημαντικοί και που θα είναι τα οχήματα αυτή τη νέα γεωργία, αυτού του νέου γεωργικού μοντέλου που χρειαζόμαστε και τέλο, Δεν θα τα κάνουμε όλα αυτά εάν δεν εμπλέξουμε και τις πόλεις ε, το αστικό ιστό σε αυτή τη συζήτηση. Ε, είναι ε, μια συζήτηση για την Ευρώπη. Δεν είναι μια συζήτηση για το αν θα στηρίξουμε τη μεγάλη παραγωγή στη χή περιοχή ή χώρα. Το θέμα είναι τι θα γίνουμε εμεί στην Ευρώπη, αν συνεχίσουμε να έχουμε μια, ένα μετασχηματισμό των γεωργικών μας υποδομών και εκμεταλλεύσεων όπως στη Βραζιλία. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη που μιλούσα τόσο γρήγορα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, σας περιορίζουμε γιατί γενικά περιοριζόμαστε όλοι από το χρόνο. Προτείνω λοιπόν να κρατήσουμε το προηγούμενο σύστημα, δηλαδή 1,5 λεπτό αναομιλητή. Ο κύριος Φλάναγκαν είναι ο πρώτος ομιλητή. Σας ακούμε. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ε, μία σύντομη ερώτηση σε σχέση με τις εμπορικές ε, συμφωνίες. Τι τύπα, Μερκοσούρ ε, και τα λοιπά και ΣΕΣΑ. Πιστεύετε ότι αυτά που, με βάση αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμή θα επιδεινωθεί η κατάσταση αν περάσουν αυτέ οι εμπορικέ συμφωνίε ή θα βελτιωθεί για τη Γεωργία. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Η κυρία Μαγκίνε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε πολλά. Έχει πολλά στοιχεία η παρουσίαση. Κάποια στοιχεία που με ανησυχούν όμω είναι το να καθορίσουμε το μέγεθος που θα έχει στην ιδιοκτησία σου ο καθένας. Ε, Παραδείγματο χάρη, ε, το ότι είναι μικρό, μικρή αγιοργική εκμετάλλευση σε ένα κράτος μέλος, ας πούμε, στην Ιρλανδία, Φερρυπή, είναι τελείως διαφορετικό από ότι στην, ε, στον Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μπορούμε να είμαστε πολύ επιτακτικοί και να βάζουμε τα, τη μύτη μα πολύ. Επίση, η γη είναι ένα αγαθό. Επίση, οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις το λέμε ξανά και εντάξει και τις υποστηρίζουμε και τα ξανά και ξανά. Αλλά ε, ο, ο ορισμός είναι πολύ ευρύς και χωράει πολύ η ερμηνεία ας πούμε και μπορεί να έχουμε μια ρομαντική εικόνα αλλά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ε, επίσης μάλλον ε, ε, είσαστε κατά τη συνεργασία των ε, γεωργών, έτσι, των συνεταιρισμών κτλ. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει τίποτα κακό σε αυτή τη συνεργασία. Ε, με οποιοδήποτε τρόπο θεωρούν καλό. Και κάθε κράτο μέλο, ό,τι αφορά τι γεωργικέ εκμεταλλεύσει και δομέ, έχει ειδικού του κανόνε. Και στην Ιρλανδία, α πούμε, έχουμε το συνταγματικό δικαίωμα στην ατομική διοκτησία. Ε, υπάρχει, είναι θέμα των κρατών μελών δηλαδή. Εξού και η σημασία αυτής της συζήτηση Και το τελευταίο, χθες ε, συμμετείχα ε, στην ε, παγκόσμια αυτή συζήτηση για την ε, πείνα στον κόσμο. Και εκεί ακόμα υπάρχουν τεράστιες διαιρέσεις ανάμεσα στον ε, αναπτυγμένο κόσμο και αναπτυσσόμενο κόσμο για το πώς, θα, πρέπει να αναπτυχθεί η γεωργία ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και εκεί υπάρχει γενικά αυτή η μικρή γεωργία, η οικογενειακή γεωργία κτλ. Και όμω ε, πολλοί από του παρεμβαίνοντε χθε είπαν ότι υπάρχει ανάγκη και σε αυτέ τι χώρε, αναπτυσσόμενε χώρε, να έχουμε μια γεωργία πιο εμπορική. Ο κ. Νταντά, ο Αλμπέρ Ντε, ε, ζητάει συγγνώμη ε, και θα, τον, θα εκφράσω τι απόψει του. Να υπενθυμίσει ότι στην παρουσίαση που ακούσαμε ακούγονται διαφορετικά πράγματα. Αλλά στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαχείριση των ε, γεών είναι αμυγός εθνική υπόθεση. Και σε αυτή τη φάση της ε, ευρωπαϊκής οικοδόμησης και αμφισβήτησης της ευρωπαϊκής οικοδόμησης νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να καταστήσουμε αυτή την πολιτική πιο ευρωπαϊκή ας πούμε ακόμα. Ε, στο βαθμό που στις θεμελιακές συνθήκες ε, στην Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέψαμε να περιορίσουμε ας πούμε το κεφάλαιο που θα έχει ο καθένας. Το ίδιο και για την ε, Γεωργία. Σήμερα στη Γεωργία ε, υπάρχει, το φαινόμενο πούμε, των εταιριών ε, που αγοράζουν γη, α πούμε, κτλ. Και, τα λοιπά, και μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα στη γεωργία, αλλά θα πρέπει να ρυθμιστούν όλα αυτά τα προβλήματα μέσω τη ε, νομοθεσία των ε, κρατών μελών. Ο κύριο Άγνιου. Είναι πάντα ενδιαφέρον να δούμε τα ακρονίμια τα οποία βγαίνουν στι διάφορε ε, γλώσσε για τι διάφορε οργανώσει. Waffle, βάφλα. Βγαίνει η οργάνωση στα αγγλικά. Είναι επικίνδυνο όμως αυτό εδώ, η οργάνωσή σας. Γιατί εξετάζουμε το τι γίνεται με, τις, ε, με την ιδιοκτησία αγιών στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη. Όταν δημοσιεύεται η είδηση πώληση ε, γεών, η αξία τους μειώνεται κατακορύφα. Τι προτείνετε δηλαδή, κρατική διοκτησία, δημόσια διοκτησία, προ αυτήν την κατεύθυνση φαίνεται ότι πηγαίνετε. Συμφωνώ ότι οι επιδοτήσει τελικά καταλήγουν στον κάτοχο των γεών και μου προκάλεσε ενδιαφέρον το τι έγινε στην, ε, στην εκστρατεία την, ε, πριν από το δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία ότι βγήκαν και είπαν ότι τελικά αυτά τα χρήματα καλό θα ήταν να καταλήξουν στην έρευνα, στην ανάπτυξη και το καθεξής. Και την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ότι οι νέοι επιχειρηματές, οι νέοι γεωκτήμονες, πώς ε, προσεγγίζουν ενδεχόμενες συμφωνίες. Για παράδειγμα, χρειάστηκε να γίνει ο ψεκασμός και κατά πόσον ε, κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίε αυτές. Ο κ. Να δώσουμε λίγο προσοχή στο παγκόσμιο προσκήνιο τι γίνεται με τις ε, συμφωνίες ότι αφορά το γεωργικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θεωρώ ότι τα γεωργικά μας μοντέλα προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε σε άλλες χώρες και έτσι αυτό σε κάποιες περιπτώσεις καταστρέφει τις παραδοσιακές δομές των γεωργών. Διακυβεύουν τα εφιστάμενα μοντέλα. Κάτι άλλο ενδιαφέρον ότι σε πολλές περιπτώσεις θέλουμε να καταργήσουμε τους εμπορικούς ε, φραγμούς για να εξαγάγουμε τα γεωργικά μας προϊόντα ενώ εμείς έχουμε επιδοτήσει και άλλοι δεν έχουν επιδοτήσει. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό, πώς επηρεάζει αυτό τις άλλες χώρες, ε, οι οικογενειακές επιχειρήσεις τώρα. Οι οικογενειακές δομές μπορεί να μεταφερθεί αυτό το μοντέλο σε χώρες που παραδοσιακά και ιστορικά έχουν συνεταιριστικές ε, δομές όπου θεωρητικά δεν υπάρχει ιδιοκτήτης κάτοχος αλλά πολύ απλά διαφέρει και η κατάσταση και εκτός Ευρώπης ε, αυτά θα πρέπει να λεφτούν υπόψη και στην εμπορική πολιτική να μην προαγάγουμε δομές οι οποίες είναι εντελώ διαφορετικές και ουσιαστικά προωθούν την εξαγωγική γεωργία. Σας ευχαριστώ πολύ. να ρωτήσουμε κατά πόσον θέλει να πάρει το λόγο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, μικρές ερωτήσεις, γιατί ακούσαμε διάφορες ε, θέσεις μεταξύ των οποίων ότι οι γεωργοί δεν θα πρέπει να δεσμεύονται από τις συγκεκριμένε εκτάσεις. Θέλουμε δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει ελεύθερη επιλογή. Φυσικά να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασία των εκτάσεων, αλλά και κατοχή. Ότι η ιδιοκτησία μάλλον των γεών δεν είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο. Και έτσι προκύπτουν μεγάλες διαφορές, μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις στον νότο στο Δεβορά Υπάρχουν άλλες, ε, ε και φυσικά υπάρχουν και οι κλιματολογικές διαφορές που δεν επιτρέπουν τόσο μεγάλες ε, διακυμάνσεις στις επιλογές. του ίδιο ισχύει και στην Ανατολική Ευρώπη, όπου έχουμε το κλωριδοδότημα του κομμουνισμού με υψηλή συγκέντρωση κοινωνική και κοινή ιδιοκτησία των γεών 15% μόνο των γεών είναι σε χέρια ιδιωτών. Η διαχείριση και η αντιμετώπιση των γεών ασφαλώς αποτελεί ζήτημα αρμοδιότητας των κρατών μελών. Και υπάρχουν λύσεις οι οποίες προτιμούνται από τα παλαιά κρατημέλη, όπως είναι για παράδειγμα η Γαλλία. Και πολύ απλά δεν μπορεί να ισχύει ανεξέλεκτα η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων. Θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός. Το θέμα λοιπόν αυτό θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε την περαιτέρω και βάσει τον όσο μας παρουσίασε η κυρία Νόχιλ στην έκθεση της, σημαντική έκθεση. Σε τελική ανάλυση το ερώτημα είναι κατά πόσον σε ε, επίπεδο θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και είμαστε ανταγωνιστικοί. Μήπως η συγκέντρωση αποτελεί ένα είδος άμυνας, ένα είδος ε, εξουδετερώσης του ανταγωνισμού. Φυσικά υπάρχει και το ζήτημα των επιδοτήσεων, των ενισχύσεων. Και εδώ θα πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ διαφορετικών επιπέδων. Όσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση, τόσο πιο μικρή είναι η επιδότηση, η ενίσχυση. Αλλά τίθεται και το θέμα της παραγωγής. Τι παραγωγή γίνεται ανά εκτάριο, ίσως αυτό οδηγεί σε μια κάποια απλοποίηση, δεν λέω. Αλλά οι μικρέ επιχειρήσεις ε, έχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα. Αλλά εμεί θα πρέπει να τοποθετηθούμε σε διεθνέ επίπεδα. <coughs> γιατί λειτουργούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Πώς όλα αυτά λοιπόν μπορούν να συγκυραστούν. Ίσως η Κομισιόν θα ήθελε να πάρει το λόγο για να απαντήσει. Αλλά πρώτα ο κύριος ε, μας. Όλες οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που διαπραγματεύεται η Ευρώπη ε, έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για την παγκόσμια γεωργική παραγωγή και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε τώρα προτού γίναν υπέρβλητα τα παγκόσμια προβλήματα. Οι συμφωνίε εταιρική εμπορική σχέση με διάφορε αφρικανικέ χώρε που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση έχουν καταστροφικά αποτελέσματα, όπω είπατε και εσεί, για την εξέλιξη τη γεωργία στην Αφρική, σε αφρικανικέ χώρε κυρίω. προωθούμε το λεσεφέρ το ελεύθερο εμπόριο το, ε, και δημιουργούμε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση σε ε, παγκόσμιο επίπεδο. Δεν χρειάζεται τώρα να επεκταθώ. Ξέρετε ότι είναι δεινή η κατάσταση. Αλλά θα κάναμε λοιπόν ε, να προβληματιστούμε για αυτά τα ζητήματα. Για τον προσδιορισμό του μεγέθου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μου είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε ούτε καν σε εθνικό επίπεδο να το κάνουμε. Είπε κάποιο σήμερα το πρωί ότι το μέγεθο πρέπει να αποφασίζει σε τοπικό επίπεδο σε σχέση με τα σχέδια που υπάρχουν, ε, τι δυνατότητε που υπάρχουν ε, στον τόπιο πληθυσμό και θα υπάρξει διακύμανση. Δεν μπορούμε να ισχύουν τα ίδια, είτε μιλάμε για την κεντρική Γαλλία, είτε για τη Σουηδία, για την Κροατία. Εξυπακούν ότι είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Ε, τώρα, για την οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση, φυσικά θα πρέπει να είμαστε ακριβέστεροι ε, και πιο συγκεκριμένοι η μεγιστοποίηση της οικονομικής επένδυσης σίγουρα δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος ενός μικρού γεωργού. Δεν είναι καπιταλιστής. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση αφενός και αφετέρου την εταιρεία παραγωγό. Ε, τι να σας πω, αν ε, ε, δεν το κρίνω. Άμα ήμουν αμέτωχος θα ήθελα μερίσματα, όσο το δυνατόν υψηλότερα γίνεται. Σε επενδύσεις στην Κίνα, στην Αφρική, άμα είναι μεγαλύτερες οι επιδόσεις, τι με νοιάζει που είναι κινητικό το κεφάλαιο. Όμως αυτή η κινητικότητα του κεφαλαίου καταστρέφει τι εγχώρες δυνατότητες σε πολλά κράτη-μέλη. Κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Δεν είναι ο στόχο να κάνουμε ιδεολογικού τύπου συζητήσει ε, για τα δικαιώματα, για τα ιδιοκτησιακά. Το θέμα είναι να είναι βιώσιμη κατάσταση που φτιάχνουμε σε κοινωνικό επίπεδο, να ε, υπερπηδήσουμε τις αντιφάσεις που υπάρχουν, να τι συμφιλειώσουμε και σε ιδιοκτησιακό επίπεδο και σε επίπεδο εκμισθώματος ε, να είναι βιώσιμη κατάσταση. Το 46 στη Γαλλία ελήφθησαν αποφάσεις ε, που ε, μετά από δεκαετίες αγώνα μας οδήγησαν σε μια κατάσταση όπου οι γεωργοί είχαν τη δυνατότητα να συνοηθούν μεταξύ τους και να εργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση όπως και η υπόλοιπη Γαλλία, οι υπόλοιποι τομείς. Δεν μιλάμε τώρα για απαλωτρίωση ε, γεών, ε, δεν είναι αυτός ο στόχος μας, ε, αλλά χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό σύμφωνο για την γεωργία και έχουμε πάρα πολλούς ανέργους στην Ευρώπη, έχουμε προβλήματα εκ και από βιομηχάνησης. Χρειάζεται λοιπόν προστασία και των εδαφών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, χρειάζεται μεγαλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στις περιοχές. Αυτά κάναμε δεκαετία του 60 και επιβιώσαμε. Λοιπόν, με τις ανταλλαγές αυτές ε, που κάνουμε εδώ, τι είναι το σημαντικό. Ε, δεν ε, κάναμε σημαντικές ανακαλύψεις, όμως ένα σημαντικό και εκτιμένο του Παγκοσμίου Φόρουμ είναι ότι επανήλθε στον πυρήνα της συζήτησης ακριβώς αυτή η απελευθέρωση των ε, ανταλλαγών. Γιατί δεν μιλάμε για ε, παραδοσιακά αγαθά και αυτό ακριβώς οδηγεί σε αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται να παραθέσω οικονομολόγους. Ο Πουλανί αυτά είπε μετά την ε, κρίση του 1929 και αυτό ακριβώς θα πρέπει να επιδιώξουμε και είναι και το διακύβευμα των μελλοντικών συζητήσεων. Δεν θα είναι απλά τα πράγματα όμως. Πρέπει να αμφισβητήσουμε τους πυλώνες ακόμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν διαπιστώσουμε ότι είναι ε, ε, παροχημένες οι επιλογές μας και δεν μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα αρρώδινο και κυρίως ειρηνικό μέλλον. Θα σταματήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μίσελ Μερλέ. Πραγματικά εμπλουτίσατε τις ε, συζητήσεις μας ε, με τις παρουσιάσεις σας ε, και η κυρία Νόιχελ σίγουρα σίγουρα θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει πολλές από τις ιδέες σας και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε γενικότερα για τα μέλη της Επιτροπής μας συνεχίζουμε Ε, ε, ε, είναι εξαιρετικά περίπλοκο και δύσκολο το ζήτημα. Σίγουρα θα επανέλθουμε στο μέλλον. Πολάκης. Θα κλείσουμε όμως προς το παρόν αυτή τη συζήτηση και περνάμε στο επόμενο σημείο. Θα πρέπει να τοποθετηθεί η Επιτροπή μας για το επόμενο θέμα, την έκθεση του κυρίου Νταντά. Ε, έχουμε αυτή την έκθεση από την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. είναι... Ο Τσάνι είναι ο εισηγητής της ΕΚΟΝ και για μας, για την γνωμοδότησή μας, ο κύριος Νταντά. Παρακαλώ, κύριε Νταντά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να χαιρετήσω και εγώ τον εισηγητή που είναι καθήλυνα αρμόδιος ε, για αυτό το θέμα και που είναι παρόν σήμερα. Ε, είναι προχωρημένη η ώρα, θα είμαι σύντομο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει κάθε χρόνο μία έκθεση για την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού και η συντονιστές ε, αποφάσισαν η Επιτροπή Γεωργίας μετά την, τα όσα συνέβησαν ε, στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ να ετοιμάσει μια γνωμοδότηση για αυτό το θέμα. Από τη στιγμή της ίδρυσης της ε, κοινή αγοράς η γεωργική αγορά έχει ιδιαίτερη θέση και ο νομοθέτης και, που ήταν το Συμβούλιο εκείνη την εποχή ε, μέσω της κοινή οργάνωσης αγοράς να δώσει ένα ειδικό καθεστώς στη γεωργία. Το σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο σας ετοίμασα είναι πολύ λακωνικό και θα το τροποποιήσετε όπως επιθυμείτε αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ προτείνω τρία επιπλέον σημεία υπομορφή τροπολογίας το θέμα της εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού σε περίοδους κρίσης, να ετοιμάσουμε, να ε, ε, μιλήσουμε για τον τομέα του βοήου και της ε, ζάχαρης, να το συμπληρώσουμε επίσης, τι γίνεται με τους διανομείς, και τι γίνεται η αντιδιαστολή ανάμεσα στους διεθνείς διανομείς και τους εθνικούς διανομείς; Ε, εμείς μπερδεύουμε το δικαίωμα ανταγωνισμού, τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Αυτά τα τρία θέματα νομίζω ότι θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε και να βάλουμε διαχωριστικές γραμμές. Υπάρχει μια άλλη έκθεση η οποία ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή για τις αθέμητες πρακτικές. Η κυρία Μαγκίνες ε, δούλεψε πολύ πάνω σε αυτό το θέμα. Ξέρω ότι η Task Force η οποία θα συναντηθεί μαζί μας τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο αφού παρουσιάσει ε, την έκθεσή της στην Κομισιόν θα κάνει προτάσεις για το θέμα αυτό. Επομένως είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει θέση και για αυτό το θέμα πριν, η Task Force κάνει τις προτάσεις της. Θέλω να τονίσω δύο ή τρία σημεία. Στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2013 είχαμε τονίσει ούτω ώστε να υπάρχουν μία σειρά από ε, παρεκκλήσεις ε, σαφείς στο δίκαιο ανταγωνισμού και διαπιστώνουμε ότι η έλλειψη σε ό,τι αφορά την εμβέλεια αυτών των ε, παρεκκλήσεων και την εφαρμογή τους από τις δημόσιες αρχές περιορίζει την ισχύ τους στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκρινίσουμε τα πράγματα, να τα καταστήσουμε ευκρινή για τους μη επαΐοντες που είναι οι γεωργοί και οι συνεταιρισμοί τους. Θα πρέπει λοιπόν επίσης να προχωρήσουμε, να δούμε τις ε, οι ιδιαιτερότητες της ε, γεωργίας σε σχέση με το δίκαιο του αγωνισμού, το θέμα της ε, δυσπόλουσας θέσης και το θέμα της σχετικής ή συναφούς αγοράς. Σήμερα έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση ε, προηγουμένως σε πρώτερη φάση στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού το υπενθυμίζει επίσης συχνά ότι έχουμε συμμαχίες που δημιουργούνται στη φάση του μετασχηματισμού με μεγάλο επιχειρήσεις, μακροεπιχειρήσεις, θα πρέπει οι γεωργοί να πάρουν θέση, να οργανωθούν χωρίς να έχουν τη δαμόκλειο σπάθη πάνω το κεφάλι τους. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι στα πλαίσια της κρίσης του γάλακτος, η Κομισιόν ε, για πρώτη φορά ε, έθεσε σε εφαρμογή το άρθρο 222 ε, για να παρεκκλίνουμε ε, από το δίκαιο ανταγωνισμού. Ε, αυτή, αυτή η παρέκκληση σε περίοδο, σε περίοδο κρίσης είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να την αναλύσουμε με προσοχή και μπορεί να υπάρξουν νέες προσαρμογές από την Κομισιόν ε, στο δίκαιο ανταγωνισμού που θα εφαρμοστούν. Ε, αυτό εφαρμόστηκε, το άρθρο 222 εφαρμόστηκε για την κρίση του γάλακτος. Έτσι. Επίσης, η αλυσίδα ε, ανεφοδιασμού σε τρόφιμα. Ε, η κρίκη σε αυτή την αλυσίδα είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα η έκθεση που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο της κυρίας Μαγκίνες να μην είναι το τέλος, να υπάρξει συνέχεια και η Κομισιόν και οι Επίτροποι να ακούσουν το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Επίσης, θεωρώ ότι η σωρευτική επίπτωση της συγκέντρωσης της διανομής σε εθνικό επίπεδο και η αυξανόμενη ανάπτυξη συμμαχιών μεγάλων διανομέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αναλυθεί από την Επιτροπή και από τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού. Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τα βασικά ε, σημεία της εκθεσής μου. Να υπενθυμίσω ότι το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σφιχτό, πολύ πιεστικό, γιατί η Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή θα αποφανθεί στις 5 Δεκεμβρίου. Η δική μας Επιτροπή ε, θα γνωμοδοτήσει απλώς και θα αποφανθεί στις 29 Νοεμβρίου. Θα είναι πολύ δύσκολο για την Αρμόδια Επιτροπή να λάβει υπόψη τις τροπολογίες μας, αυτή στιγμή ψηφιστούν οι συμβαστικές δηλαδή τροπολογίε ψηφιστούν και να τις ενσωματώσει στο κείμενο τη. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, μέσω επαφών τις επόμενες ώρες μεταξύ αδίσκιωδών δηλαδή, ε, εισηγητών και εισηγητών να μπορέσουμε να καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες δικές μας ούτω ώστε να μπουν απευθεία ε, στο κείμενο τη καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, ούτω ώστε να τι λάβουν υπόψη και οι σκιώδεις και ο, σκιώ, και ο εισηγητής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Για ένα μισή λεπτό μόνο να πάρετε το λόγο. Κύριε Τεκάστρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θέλω να τονίσω ότι η δουλειά του Μισελ Νταοντάν είναι πάρα πολύ λεπτή δουλειά, πάρα πολύ σημαντική δουλειά και αφορά το βασικό έργο της Επιτροπής μας και στην έκθεση της κυρίας Μακίνης ασχοληθήκαμε με το θέμα του θεμητού ανταγωνισμού στο εσωτερικό της Γεωργίας με είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευτυχώς ο γενικός συγητής του θέματος αυτού είναι ο Τίμπορ Τζάνι, που είναι συνάδελφος και κατά γνώμη θα μπορέσει να λάβει υπόψη τη δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ. Δηλαδή μέσω του Μισελ ας πούμε. Και σε ευχαριστώ Μισελ γιατί όλα τα πράγματα που είπες είναι ο καρπός μιας δουλειάς που κάναμε μαζί από την αρχή. Σε ευχαριστώ που καταφέρνεις με αυτά τα λόγια σου, ε, παρά το γεγονός ότι έχουμε αυτό το προβληματικό χρονοδιάγραμμα, να περάσεις και τις απόψεις της Επιτροπής Γεωργίας. Σας ευχαριστώ, λέγει ο Πρόεδρος. Το πρόβλημα λοιπόν, ξέρετε, είναι ότι είναι μάλλον γνωστό στου συζητητέ. Ο κ. Μπέιλτερ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και το Σκιώδη. Να πω ότι ο Σκιώδη ε, ε, ε, εισηγητή του ECR είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον συνάδελφο Ντάντα για την ισορροπημένη του αυτή έκθεση και εργασία. Θεωρώ ότι κοιτώντα την Task Force έχουμε να αντιπαρατηρήσουμε ότι η συλλογική δράση αποτελεί αρμοδιότητα τη Task Force σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες περιμένουμε να καταθέσει προτάσεις η, η Task Force για τα ζητήματα αυτά. Και επίσης όλα αυτά θα πρέπει να λεφτούν υπόψη στα πλαίσια της βιωσιμότητας και τα κοινωνικά, τα κοινωνικά ζητήματα είναι σημαντικά. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία με τον εισηγητή, δεδομένου και του χρονικού για προγράμματο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε κυρία Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον κύριο Νταντάν για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, που είναι πάρα πολύ καλή και την οποία υποστηρίζει στις γενικέ γραμμές σε ό,τι αφορά την, το σημείο 4, την δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι Υπάρχει έκθεση από το Ιρμανικό Υπουργείο για τα Καρτέλ σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Και θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ θετικό το γεγονό ότι συμπεριλαμβάνεται και η έκθεση τη κυρία Μαγκίνε για τι αθέμητε πρακτικέ. Ένα πράγμα είναι σαφέ, ότι υπάρχει μία έλλειψη ισορροπία σε ό,τι αφορά τι ε, γεωργικέ, του γεωργικού συνεταιρισμού και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην γίνονται τέτοιε συμφωνίε για καλύτερε τιμέ και το καθεξή. Και θεωρώ ότι μπορούμε να κινηθούμε και πολύ περαιτέρω από αυτά που προτείνει ο συνάδελφο Ντάντα. Νομίζω ότι το τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο δημιουργεί προβλήματα τίθεται και θέματα Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των συνεταιρισμών ή εθελοντικές πρωτοβουλίες. Τις καλωσορίζουμε. Αλλά ουσιαστικά πολύ μεγάλε ομάδε ε, γεωργών δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Ε, προς την κατεύθυνση λοιπόν αυτή θα καταθέσω τροπολογίε. Μάλιστα λέει ο Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Όλα καλά λοιπόν. Αν ε, η Άλντε μιλάει έτσι είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Ο κ. Λουαζό. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε σε ό,τι αφορά το σημείο 1 και 2 του θέματο, Είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση όντω επιτρέψε τη δημιουργία μια πολιτική για την προώθηση της ελεύθερης, ε, του ελεύθερου ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά τη διακύβευση τώρα των θέσεων εργασία. αυτό έβαλε τους γεωργούς σε μια μοιραία ε, σε ένα μοιραίο φαύλο κύκλο ανταγωνισμού. Και όπως ξέρετε, δεν έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια προ την κατεύθυνση αυτή. Η λύση θεωρώ ότι θα ήταν να μπει ένα τέλο ε, στον ανταγωνισμό αυτό, εφαρμόζοντας μία πολιτική συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για ανταλλαγή προϊόντων τα οποία πραγματικά χρειάζεται το κάθε κράτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρος Μακίνες, ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε και να υποστηρίξω εν συντομία το έργο του κ. Νταντάν γιατί στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ήσασταν πραγματικά εμείνατε σε θέματα πολιτικής ανταγωνισμού και το πετύχατε αυτό με την γνωμοτότηση αυτή και κατά δεύτερον νομίζω ότι θα πρέπει να στείλουμε και επιστολή στέλνουμε μάλλον επιστολές στον Επίτροπο ένα θέμα που δεν έχουμε δείξει επαρκώς όμως είναι το θέμα της ε, παροχής από τις εταιρείε, της προσφοράς από τις εταιρείε ε, και τους μεγάλους ομίλους και το τι συνέπειες έχει η διαδικασία συγχωνεύσεων στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας. Θα πρέπει να το δείξουμε αυτό προς τον Επιτροπά. Επίσης, συγκέντρωση στον τομέα παραγωγής κρέατος στην Ιρλανδία. Πέρασε η σχετική ρύθμιση από την Επιτρόπο και αποφάνθηκε ότι δεν είναι πρόκειτο για θέμα ανταγωνισμού και δίκαιο ανταγωνισμού. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αποτελεί αυτό θέμα ανταγωνισμού. Το ίδιο πιστεύουν και η παραγωγή μας στην Ιρλανδία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία με το έργο σας, λοιπόν, γιατί θα χρειαστείτε. Είναι δύσκολο το έργο σας. Ευχαριστώ, και ο Σας ευχαριστώ. Και ο κ. έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τοντάμ. Σας ευχαριστούμε που γράψατε αυτή την έκθεση. Είναι ισχυρό το μήνυμα που θέλετε να περάσετε και είναι σημαντικό το ζήτημα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Και θέλω να συζητήσω με όλους ποιος είναι ο καλύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος να αυξήσουμε την διαπραγματευτική δύναμη του πρωτογενούς ε, τομέα των ε, γεωργών. Ε. Και γιατί το ρωτάω, διότι προβλέπονται εξαιρέσει για τα γαλακτοκομικά παραδείγματο χάρη ή βάση του άρθρου 222. Όμως δεν μπορούν οι γεωργοί να τα χρησιμοποιήσουν, να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εξαιρέσεις. Λοιπόν, εάν τους δώσουμε δυνατότητα να αποκλίνουν από το δίκαιο ανταγωνισμό, θα πρέπει λοιπόν και ο πρωτογενής τομέας να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία να τη χρησιμοποιήσει. Γιατί οι άλλοι τομεί μπορούν να μας πούνε γιατί έχει η Γεωργία αυτές τις εξαιρέσει και εμεί όχι. Και γιατί δεν τις χρησιμοποιούν τι εξαιρέσει οι Γεωργοί. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Είναι σημαντικό στοιχείο. Και δεύτερον, σε σχέση με τα συμπεράσματά σας στην έκθεση. Υπάρχει και η Task Force για την γεωργική αγορά ε, και τα, οι τη. Ε, θα ήθελα και αυτό να ληφθεί υπόψη. αν μπορείτε να τις ενσωματώσετε στην ε, γνωμοδότησή σας. Και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο τομέας της Λιανικής, αλλά και οι προμηθευτές, γιατί έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ σε σχέση με τον πρωτογενή. Έχουν καλύτερη θέση στο δίκαιο ανταγωνισμού ή ο πρωτογενής τομέας έχει αυτές τις δυνατότητες αλλά δεν λειτουργεί αποτελεσματικά ούτως ώστε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του ισχύ. Είναι άνηση η ε, θέση που, έχουν, ε, που έχει πρωτογενή στο μέσο ολόκληρη την αλυσίδα. Με ευχαριστούμε. Ο κύριος Φλάνιγεν. Ε, Θέλω να συγχαρώ τον Μίσελ για τη δουλειά του. Λέει πολλά σωστά πράγματα. Το ίδιο και η κυρία Μαγκίνες στην προηγούμενη έκθεση. Φαίνεται όμως ότι η δεξιά κάνει αυτό και η αριστερά η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ακολουθούν την ε, αντίθετη κατεύθυνση και ε, υπονομεύουν τις αποφάσεις ε, των αρχών ανταγωνισμού ε, της συγχώνευσης ε, της Γενικής Δηλαδή και σχεδόν 30% του τομέα κατέχουν και 50% της ικανότητας απόδοσης για, τα εντόστια για την διάθεση των εντοστίων. Πώς να ανταγωνιστούν λοιπόν οι γεωργοί. Εκεί αναφέρεται ότι το μέγιστο μερίδιο της αγοράς για τις ενώσεις παραγωγών είναι 15% καταλαβαίνετε. Είναι, μιλάμε για ε, ε, ένα αστείο διότι δεν... Ε, είμαστε σοβαροί, θέλουμε να κάνουμε ε, κάτι για τον ανταγωνισμό. Σοβαρότατο το πλήγμα κατά τη Ιρλανδία την περασμένη εβδομάδα και μας λέτε όλα καλά. Ε, τότε τι κάνουμε εδώ πέρα. Μήνες ολόκληρο, γράφουμε επιστολές ε, και ε, ασχολούμαστε με τα γραμματάκια θα μπει τι θα μπει ε, και εσείς ε, κάνετε τέτοια εξόφθαλμα πράγματα. Χειροτερεύει ε, η κατάσταση. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε κύριος Άγνιο. δεν... Ε, φοβάμαι τους. Ε, δεν, ε, από τις προηγούμενες ομιλητές δεν μου δημιουργούν τράκα, αλλά αυτή τη στιγμή ο Φλάνναγκαν το κατάφερε. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση, μια, όχι έκθεση, μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Οικών. Και οι γνωμοδοτήσεις, ξέρετε, γενικά δεν βγάζουν ούτε το χαρτί που χρησιμοποιούν. Ας μην το αρνούμαστε. Αυτό που με ανησυχεί είναι το τι γνωρίζει η Επιτροπή Οίκων για το Ηνωμένο Βασίλειο και για τα παραγωγή λαχανικών, δεν θέλω πραγματικά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να δυσκόλεψει περαιτέρω τα πράγματα, γιατί έχει αρχίσει να σημειώνεται κάποια πρόοδο και τα τέσκο τα σούπερ μάρκετ μα. Έχουν αλλάξει πολύ τον τρόπο που λειτουργούν. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι έχουν γονατίσει κιόλα ε, σε, ό,τι αφορά την απλοποίηση. Ένα τα θέματα που αναφέρονται. Θα ήθελα να κοιτάξουμε λοιπόν τι συμβαίνει ήδη και ποια κατάσταση διαμορφώνεται. Ο αγρότης παίρνει τα χρήματα των προλογημένων για να μειώσει την παραγωγή γάλακτος εκ παραλίλου. Ο ίδιος αγρότης παίρνει χρήματα από τον αγοραστή του γάλακτος, από ένα συνεταιρισμό, για να παράγει πιο πολύ. Τέτοιες καταστάσεις λοιπόν προκαλεί η υπερβολική παρέμβαση στις αγορές. Ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Νταντά για αυτή την έκθεση. Είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό να δώσουμε και δυτική μας γνώμη, ούτως ώστε να επηρεάσουμε την κατάσταση τουλάχιστον στην ε, Ήπεθρο. Γιατί σήμερα είναι σαφέ ότι δεν υπάρχει δίκαιο ανταγωνισμό. Στι βαλτικέ χώρε, Φερρυπίν, στη Λιθουανία, τα τελευταία χρόνια, το 1 τρίτο των γαλακτοπαραγωγών πτώχευσαν. Επειδή δεν υπάρχει ισοτιμία μεταξύ των διαφόρων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, διάφορες ε, εκμεταλλεύσεις πτωχεύουν. Το εισόδημα των εισαγωγών, των ε, γεωργών, εξαρτάται από τις τιμές και από τις ενισχύσεις. Και υπάρχουν τεράστιες διαφορές από κράτος σε κράτος μέλος. Είναι πολύ δύσκολο να ανταγωνιστούν οι γεωργοί δίκαια ο ένας τον άλλον. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα δίκαιο σύστημα πληρωμής και μια δίκαιη αλυσίδα ανεφοδιασμού. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει η γεωργία μας ανταγωνιστική. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο στον εισηγητή της Επιτροπής ΕΚΟΝ, ε, που ξέρει πολύ καλά το πρόβλημα. Είσαστε και υπουργό στη χώρα σας. Σας δίνω το λόγο, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας πω ότι με πολύ ενδιαφέρον άκουσα και τις ε, θέσεις σας Ως εισηγητής για το θέμα αυτό από την εικόνα. Να ενημερώσω ότι φέτος θα ακουστούν οι ενστάσεις σε ό,τι αφορά την Ιρλανδία και άκουσα τα σχόλιά σας. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να μου τα εξηγήσετε λίγο καλύτερα όλα αυτά. Γιατί στην τελική ανάλυση η δουλειά μου θα είναι να συνενώσω όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις σε ένα ενιαίο έγγραφο. Χαίρομαι λοιπόν που η Επιτροπή Οικονομικών ε, συγγνώμη, γεωργική ανάπτυξη και ο φίλο μα, ο κ. Ντάντα, δαπάνησε τόσο πολύ ενέργεια για να δημορφώσει με θετικό τρόπο την κατάσταση αυτή. Και κατανοώ. Την ισορροπία σε ό,τι αφορά τα σχόλια τα οποία μοιράστηκε μαζί μας. Δύο στοιχεία λοιπόν θα ήθελα να τονίσω. Καταρχάς ότι η έκθεση αυτή θα αναγνωρίσει ότι η γεωργία δεν μπορεί να μπει σε ένα καζάνι με οποιοδήποτε άλλο τομέα. Γιατί εδώ μιλάμε για θέματα βιολογίας, ασφάλειας του καταναλωτή. Όλα αυτά τα θέματα, καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο σημαντικά από οποιαδήποτε άλλη παραφιλολογία για την ε, ανταγωνισμό. Κάτι άλλο που ήθελα να θέξω και αυτό θα ήθελα να ζητήσω να το εξετάσει και η Επιτροπή σας. Την εβδομάδα αυτή που ε, απονεμήθηκαν και τα βραβεία Νόμπελ έλαβαν δύο επιστήμονες ε, ένα βραβείο Νόμπελ και εδώ συνειδητοποιούμε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία στα οικονομικά ζητήματα. Συνεργασία, όχι ανταγωνισμός. Αυτή την ε, νοοτροπία θα έπρεπε να προωθηθείτε, να προωθήσει η έκθεση αυτή τώρα που γνωρίζουμε και πώς ε, δόθηκαν τα βραβεία Νόμπελ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ας γίνει αυτό, δεν το ελπίζουμε. Μπορούμε να ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ο κύριος Πόλης Ισά. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ. μη. Ε, βουλευτές, ε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε που επανειλημμένα μας προσκαλείτε για να υποβάλουμε αναφορά σε σχέση με τις πρώτες εργασίες της ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ ανταγωνισμού. Θα θέλαμε να συνεχιστεί ε, αυτός ο διάλογος επίσημα ή επίσημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ζητήματα που θέσατε, όχι μόνο για σας αλλά και για μας. Πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Νταντάν και τα επακόλουθα σχόλια μας βρίσκονται σύμφωνος. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική ισχύ και τη θέση των γεωργών στην Ευρώπη. Ε, ο νέος αρός βουλευτής ε, έθεσε ακριβώς αυτό το κέριο ερώτημα. Τι είμαστε αντίθετοι. Το 2013 με την μεταρρύθμιση κάναμε σημαντικότατο βήμα σε σχέση με τις αποκλήσεις από το δίκαιο ανταγωνισμού που είναι υποφελής για το γεωργικό τομέα και για τους γεωργούς. Πιο συγκεκριμένα, εξαιρέσεις ε, που αποτελούν και κίνητρο συνεργασίας ε, των ε, γεωργών. Ο κύριος Τσάνη αυτό είπε στο τέλος. Και για το πακέτο των γαλακτοκομικών προϊόντων, οι εξαιρέσει και η έγκριση συμφωνιών ποσοστώσεων δεν βοηθάει τους γεωργούς και σίγουρα δεν εξυπηρετεί πολλούς στόχους κοινή γεωργικής πολιτικής μακροπρόθεσμα. Όντως δεν είναι υποφελής για τους γεωργούς. Ποιο είδους εξαιρέσει θα τους βοηθούσαν ε, λοιπόν. Ερωτάτε επαναλαμβάνω ότι τα, τα σωστά ε, βήματα έγιναν ε, και το λέω με ταπεινοφροσύνη το 2008 σε κάποιους τομείς οι γεωργοί μπορούν να εξαιρεθούν από τους γενικούς κανόνες ανταγωνισμού αν επιδιώξουν τη συνεργασία, πέρα δηλαδή από την προσπάθεια να καθορίσουν τις τιμές, αν σχεδιάσουν κοινή παραγωγή ή αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη κοινή δραστηριότητα. Με τα χαράς να επεκταθώ. Θέλω όμως ε, πρώτα απ' όλα ε, να σχολιάσω τη συγχώνευση των σφαγίων ε, στην Ιρλανδία που ενέκρινε πριν από λίγες μέρες ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. στο τελευταίο έξι μήνες είδαμε, εξετάσαμε την κατάσταση και όταν φτιάχνουν συνεταιρισμούς οι γεωργοί και συγχωνεύονται, οι αρχές ανταγωνισμού ε, και η Επιτροπή ενέκρινε πολύ ψηλότερα επίπεδα συγκεντρωτισμού σε σχέση με τα σφαγεία ε, στην Ιρλανδία. Σίγουρα λειτουργούμε ε, με δικαιοσύνη και δεν είναι προσπαθούμε να δυσκολεύσουμε τη ζωή των γεωργών σε σχέση με άλλους τομείς. Είναι ξεκάθαρα, προκύψει άθαρα αυτό από τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έγινε και ένα σχόλιο, πολύ σοφά, σε σχέση ε, με τη σχέση των ε, κανόνων ανταγωνισμού και των πρακτικών ε, θεμητών όρων ανταγωνισμού. Ε, υπάρχει καλός και κακός ανταγωνισμός. Προσέξτε, και ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχουν αθέμετοι όροι ανταγωνισμού. Δεν ε, έχουμε τέτοιο θέμα. Δεν προστατεύουμε τέτοιου αθέμητου όρου εάν δεν πληρώνονται τα τιμολόγια ή πληρώνονται με καθυστέρηση τα τιμολόγια ή οτιδήποτε άλλο που πλήττει του γεωργού. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο αποτελεσματικό ανταγωνισμό εξυπηρετεί μακρόπνοα τα, συμφέρ τα, τους στόχους της ε, κοινής γεωργικής πολιτικής και τα συμφέροντα των γεωργών, διότι η μακροπρόθεσμη, η βιώσιμη γεωργία, μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να επιβιώσει αν καταρρεύσουν οι γεωργοί. Σε περίπτωση που εξετάζεται το ενδεχόμενο περαιτέρω εξαιρέσεων για τον γεωργικό τομέα, που είναι ένα ε, τομέα με ιδιαιτερότητε, ε, αυτού θα συμφωνήσουμε, να έχετε κατά νου ότι δεν πρέπει να είναι απλές εξαιρέσεις που επιτρέπουν ε, καθορισμό τιμών, αλλά να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία ανάμεσά τους με συνεταιρισμούς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και νομίζω ε, θα ε, υποφεληθούν όλοι μακροπρόθεσμα από αυτό. Σας ευχαριστώ και εδώ είμαι αν έχετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας την ιδιαιτερότητα της γεωργικής αγοράς στην πολιτική ανταγωνισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Χαίρομαι που είπατε ότι κινούμαστε προς σωστή κατεύθυνση και ότι είμαστε στο ίδιο μήκο κύματος ε, εσείς και εμείς. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στο Γιώργο Νταντάν για να μας πει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, για, την, για τα όσα είπατε. Ε, με αυτόν τον, τρό, ε, τον τρόπο αυτά που λέω εγώ δεν, μοιάζουν, δεν με σκιάχτρο ας πούμε για τη Γενική Διαθήση Ανταγωνισμού γιατί ξέρετε ότι μερικές φορές ε, η Γεωργία ας πούμε φοβίζει μέσα υπηρεσίες της Κομισιόν. Ε, έλαβα υπόψη μου κάποια από τα πράγματα που άκουσα. Ε, θέλω να κάνω ανταλλαγές ε, το θέμα είναι ότι εγώ ε, με τον πρόεδρο της Task Force, ε, επειδή μένουμε μακριά, δεν είναι τόσο εύκολο να επικοινωνήσουμε. Θέλω να το κάνω όμως. Επίσης, εάν οι προτάσεις μου ενόχλησαν τον Βρετανό ε, νομοθέτη, ε, από ό,τι ξέρω δεν θα μείνετε και για πολύ, επομένως ε, ας, ανεχτούμε οι μεν τους δε για το λίγο χρόνο που μας μένει κοινή ζωής. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε γεωργικά καρτέλ, γεωργικέ συμπράξει. Θέλουμε να εξορροπήσουμε τις σχέσεις. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να φτιάξουμε καρτέλ ε, παράνομα ή νόμιμα γεωργικών παραγωγών. Ε, θέλουμε μία σαφή, ξεκάθαρη αγορά, όπου καθένας θα έχει τη θέση του, όπου δεν θα πλουτίζουν κάποιοι βάρος κάποιοι άλλων και δυστυχώς αυτοί που είναι τα θύματα είναι συχνά η παραγωγή. Πρόεδρος, πολύ ωραία. Έχετε μέχρι τις 18 Οκτωβρίου για να καταθέσετε τις τροπολογίες σας. Κύριε Φλάναγκαν. Μπορείτε να θέσετε απευθείας το ερώτημά σας στην Κομισιόν, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Εντάξει, συμφωνείτε. Πολύ ωραία. Κύριε Νταντά, Πρόεδρε, δεδομένου του λίγου χρόνου, και κατά παρέκκληση από τους συνήθεις κανόνες να ζητήσω τους συναδέλφους να μου στείλουν τις τροπολογίες τους αν είναι ε, στα αγγλικά ε, και σε μένα μαζί με τη γραμματεία γιατί θα πρέπει ε, όσο πιο γρήγορα κινηθούμε απέναντι στην Επιτροπή ΕΚΟΝ θέλω να πω τόσο το καλύτερο τόσο πιο σίγουροι θα είμαστε θα λυθούν υπόψη οι παρατηρήσεις μας μεταξύ Τρεις και τέσσερις συνάδελφοι, 15 και 16, έχουμε μια κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών ΔΕΒΕ, ΆΓΡΙ και ε, ΕΒΙ ε, για την Διεθνή ημέρα ε, επισητιστισμού. επισητιστισμού. Λοιπόν, η συνεδρίαση αυτή θα γίνει στην αίθουσα 2Q2 από τις 3 μέχρι τις 4. Θα είναι κρίμα να μην έρθετε εσείς. Παρακαλώ οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Γεωργίας να είναι παρόντες. Θα ήταν κρίμα όλες, όλοι οι άλλοι βουλευτές να είναι παρόντες και όχι της Επιτροπής Γεωργίας. Λοιπόν, τρεις με τέσσερις, έτσι. Τώρα, κλείνει αυτή η συνεδρίαση και περνάμε συνεδρίες των συντονιστών. Ευχαριστώ κύριε Νταντά ε, και ζητώ συγγνώμη κύριε Φλάνναγκα που δεν σας άφησα να ξαναμιλήσετε.